Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω όλους στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το σεμινάριό μας, το σεμινάριο δικαίου, Καλωσορίζω λοιπόν τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί βεβαίως το σεμινάριο αυτό οργανώνεται με τους εθνικούς βουλευτές. Έχουμε 21 βουλευτές από 28 εθνικά κοινοβούλια. Λαμβάνοντας υπόψη ε, τις ε, ατμοσφαιρικές και κλιματικές συνθήκες ε, που δεν είναι πάρα πολύ καλές σήμερα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα που έχουμε επιτύχει είναι πολύ ικανοποιητικό. Αυτή είναι ήδη η δεύτερη φορά που συναντιόμαστε και επομένως ε, έχουμε ξεκινήσει έναν εντατικό διάλογο ανάμεσα στις ε, αντίστοιχες ε, επιτροπές νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τα θέματα τα οποία θα μας αποσχολήσουν σήμερα είναι η οικογένεια και οι πολίτες ε, της Ευρώπης. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε από πλευράς δικαίου. Νομίζω ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί έχουμε όλο και περισσότερες διασυνοριακές υποθέσεις είτε ε, από οικογένειες ε, οι οποίες έχουν συντεθεί από διάφορες εθνικότητες ή μιας εθνικότητας που ζουν σε άλλες χώρες. Έχουμε κληρονομικό δίκαιο το οποίο γίνεται όλο και πιο περίπλοκο σε αυτήν την ολοκληρωμένη Ευρώπη και επομένως πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο για να μπορέσει να διευκολυνθεί το θέμα για τους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να έχουν πρακτικές απαντήσεις και όχι μόνο θεωρητικά ερωτήματα σαν αυτά τα οποία εμφανίζονται εδώ. Γι' αυτό και θα έχουμε μία σειρά από μιλητές. Θα ήθελα καταρχήν ε, να ε, χαιρετήσω την κυρία Γόλης η οποία είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συγγήτρια εδώ η οποία θα αναλάβει και μία θεματική ενότητα για να προεδρεύσει διότι κάποια στιγμή εγώ δυστυχώς θα χρειαστεί να σας εγκαταλείψω ε, θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον εκπρόσωπο της βελγικής κυβερνήσεως τον κύριο Μελχιόρ Βατλέ ο οποίος είναι πρόσωπος ε, για τα θέματα προϋπολογισμού, ε, μετακίνησης και πολιτικής ασύλου και οικογενειακής πολιτικής. Δεν μπορώ ακόμη να χαιρετήσω την κυρία Ρέντινγκ, διότι η κυρία Ρέντινγκ θα έρθει κατά τις 10 ε, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων προβλέπω ότι θα είναι λίγο καθυστερημένη στην άφηξή της και ε, υπάρχουν και πολλοί άλλοι τους οποίους θα ήθελα να χαιρετήσω και συγχρόνως όλους εσάς στους οποίους εύχομαι καλές συζητήσεις επίσης τεχνικά θέματα θα ήθελα να σας πω ότι όποιος θέλει να θέσει μία ερώτηση έχει μπροστά του ένα δελτίο το, το οποίο μπορεί να συμπληρώσει και να το δώσει εδώ στο Προεδρείο κατά τρόπον ε, ώστε να μας διευκολύνει όταν καταρτίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών παρά να χρειάζεται να κοιτάξουμε μέσα στην αίθουσα ποιος θα ήθελε να παρέμβει. Ε, έχετε πάρα πολλά έγγραφα πάνω στο τραπέζι ε, για τα διάφορα επιστημονικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες οι οποίοι μέχρι μέχρι στιγμή ε, τα έχουν καταρτήσει και ε, όντως ε, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για εξαιρετικά έγγραφα. Οπότε εφόσον ολοκλήρωσα θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γουόλης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου του Προεδρείου και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Γιάννη Μπούζεκ, θα ήθελα να σα καλωσορίσω και πάλι θερμά και να πω λίγα λόγια για το πλαίσιο της σημερινής μας συνεδρίασης. Δηλαδή για το έργο που έχει επιτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια και το έργο που ευελπιστούμε ότι με τη δική σας αρρωγή και υποστήριξη θα επιτελέσουμε και στο μέλλον προκειμένου να διευκολύνουμε κατά πολύ τις ζωές των συμπολιτών μας, των οικογένειών τους, και τι ε, δραστηριότητε γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημείο αφετηρία, κατά τη γνώμη μου, έλαβε χώρα πριν από αρκετά χρόνια, που σε μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε πει ότι σε θέματα ελεύθερης διακίνησης διαπιστώναμε ότι είναι πιο εύκολο να διακινεί κανείς εμπορεύματα, ένας εκεί πατάτες για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ότι να διακινούνται ελεύθερα οι συμπολίτε μα. Δεν μπορούσαν οι πολίτε να αξιοποιήσουν αυτό το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν, λοιπόν αυτή την πραγματικότητα. Και είπαν και οι κυβερνήσει ότι οι πολίτε έχουν το δικαίωμα τη ελεύθερη κυκλοφορία. Οπότε αυτό το θεωρούν πια δεδομένο και το απαιτούν οι συμπολίτε μα. Αν ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία, το 2009 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή να μένουν, να εργάζονται, να συνταξιοδοτούνται, να παίρνουν τη σύνταξή τους ή να φοιτούν σε άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στην πατρίδα τους δηλαδή. 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες και μάλιστα γνωρίζουμε ότι ο αριθμός αυτός όλο και αυξάνεται. Αποτέλεσμα αυτής της αυξανόμενης κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών είναι σαφές ότι ε, συνηθισμένα περιστατικά του βίου όπως ε, ε, ο γάμος, η απόκτηση παιδιών, το διαζύγιο, ο χωρισμός, ακόμη και ο θάνατος έχουν διασυνοριακές νομικές ένομες συνέπειες. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που είναι πιο ευάλωτος και το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να προσκρούσει σε περίπλοκα διασυνοριακά νομικά προβλήματα. Δυστυχώς αυτό αυτό το τελευταίο και παρά το έργο που έχουμε επιτελέσει είναι κάτι το σύνηθες. Δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά, διοικητικά και πρακτικά προσκόμματα και δυσκολίες εξαιτία των διαφορετικών νομικών μας συστημάτων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση διαζυγίου, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, τι γίνεται με τις κληρονομίες, ποιο κληρονομικό δίκαιο ισχύει. Και υπάρχουν και διασυνοριακά θέματα, επίσκεψη παιδιών πρόσβαση στα παιδιά αλλά ακόμη και η αναγνώριση, η, η ύπαρξη ε, απλών εγγράφων οικογενειακής κατάστασης είναι δύσκολη μερικές φορές. Οπότε η ζωή σε μια Ευρώπη που προωθεί την κινητικότητα δεν είναι τόσο απλή όσο θα μπορούσε ή θα όφιλε να είναι. Όλοι όσοι έχουμε τα τελευταία χρόνια ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στην Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Βέβαια, Όλοι αυτή τη στιγμή απασχολούμαστε με τα εθνικά μας δικαστικά συστήματα και την ε, περιορισμένη πρόσβαση σε, στη δικαιοσύνη εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Αλλά δεν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να προσθέσουμε άλλο ένα στρώμα περιπλοκότητας και με το διασυνοριακό χαρακτήρα, με τη διασυνοριακή διάσταση που μπορεί να εμποδίσει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν ε, διακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμένουν ή εργάζονται αλλού. Αν λοιπόν απλουστεύσουμε τα νομικά ζητήματα, τα περισσότερα νομικά ζητήματα και αν όλο και περισσότεροι πολίτες μπαίνουν στο πειρασμό να αξιοποιήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, αυτή η εσωτερική κινητικότητα ίσως δώσει ε, μία όθηση και στην οικονομική δραστηριότητα και οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη. Μην θεωρήσετε ως ε, νότα πισιοδοξία αυτά που σα είπα, γιατί μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και για την πρόοδο που έχουμε παρατηρήσει, γιατί όντω κάποια εμπόδια έχουν καταπέσει. Για παράδειγμα, υιοθετήθηκε ο κανονισμό ε, Βρυξέλλε 2 για τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων σε γαμικά ζητήματα και σε θέματα γονική ευθύνη. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και τη ε, για θέματα συντήρησης, διατροφής και μάλιστα σε πολλά κρατημέλη συνεχίζεται το έργο για θέματα διαζυγίου και κληρονομικά ζητήματα. Βέβαια, πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της διευκόλυσης της διασυνοριακής προστασίας των δικαιωμάτων γονέων και παιδιών, ενισχύοντας τη διαμεσολάβηση μεταξύ των συζύγων, να εξασφαλίσουμε αναγνώριση διεθνών αποφάσεων υιοθεσία και να αντιμετωπίσουμε ε, κάποιες νομικές δράσεις ε, ε, από άγωνα αποστήρα ζευγάρια υποκατάστατη της για παράδειγμα. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και πολλοί πολίτες τα αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν πολλά διασυνοριακά προβλήματα που αφορούν θέματα περιουσιακής κατάστασης των συζύγων, αλλά ε, γαμικών σχέσεων ή σχέσεων μεταξύ ανθρώπων που συμβιώνουν χωρίς να είναι παντρεμένοι. Υπάρχουν και θέματα οικογενειακής βίας, ακόμη και αναγκαστική γάμη, γιατί στην Ευρώπη έχουμε τέτοια εγκλήματα. Ποια είναι λοιπόν η αντίδραση των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Έχει καταστεί σαφές κατά το πρώτο έτος ε, εφαρμογής της νέας εντολής και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει βούληση και μάλιστα άνευ προηγουμένου βούληση, να θέσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες στην καρδιά των πολιτικών μας και της χάραξης της κοινωνικής στρατηγικής, ιδιαίτερα στα θέματα του αστικού δικαίου και της αστικής δικαιοσύνης. Έχουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έναρξη της θητείας της και έχουμε και την θετική απόκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επικροτεί αυτή την κατεύθυνση. Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια αντανάκλαση αυτής της αλλαγής και στη... στις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών και τα τελευταία αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου για θέματα αστικού δικαίου διαπιστώνουμε ότι δύο τρίτα, που είναι πολύ εντυπωσιακό στοιχείο, δύο τρίτα όσων ερωτήθηκαν έδωσαν την απάντηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να λάβει πρωτοβουλίες για διασυνοριακά ζητήματα οικογενειακού δικαίου. Είναι πολύ εντυπωσιακή λοιπόν αυτή η στήριξη και μας δημιουργεί την υποχρέωση να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες. Και νομίζω όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να ε, υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι αυτό το βήμα δεν ε, ε, σημαίνει εναρμόνιση. Δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί οι περισσότεροι καταγόμαστε από νοοτροπίες, από πολιτιστικές παραδόσεις, αλλά και νομικές παραδόσεις, ε, για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι. Και δεν θέλουμε που δεν είναι να διαλύσουμε ή να καταργήσουμε αυτά τα νομικά συστήματα. Απλώς θέλουμε με διάφορα συστήματα και καθεστώτα διεθνούς δικαίου να αναγνωρίσουμε τα διάφορα συστήματα που θα γίνουν συμβατά μεταξύ τους και να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων νομικών συστημάτων. Αυτό είναι ο στόχος μας για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των συμπολιτών μας που αξιοποιούν τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας και διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνας χορηγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια και το τονίζω αυτό διευρυμένες αρμοδιότητες και δυνατότητες στα θέματα αυτά προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ε, των πολιτών και των οικογενειών τους. Γι' αυτό και η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τη σχέση μας και να εντείνουμε τη συνεργασία μας στο μέλλον. Όχι βέβαια μόνο για θέματα αστικού δικαίου, αστικής δικαιοσύνης. Ε, θα πρέπει, και είναι σημαντικό για όλους μας, να αναμίξουμε και τους ε, νομομαθείς, ε, τους δικαστικούς, τα κράτη-μέλη, όλους τους ενδιαφερόμενους του κλάδου, γιατί αυτοί καθημερινά εφαρμόζουν τις πολιτικές που εμείς προσπαθούμε να επεξεργαστούμε και να θεσπίσουμε. Οπότε η ανάμειξή σας και η δική τους ανάπτυξη, ε, ανάμειξη από την αρχή είναι κέρια σημασία για να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Για μένα λοιπόν Συνιστά ιδιαίτερη χαρά η διεξαγωγή της συνδιάσκεψης αυτή σήμερα και με εντυπωσιάζει ο πλούτος της ημερήσιας διάταξης και ο όγκος των εγγράφων κάτι που προαναγγέλει μια πολύ αναβαθμισμένη συζήτηση πολύ καρποφόρα και ποιοτική και χαίρομαι που έχουμε και τον εκπρόσωπο της Βελικής Προεδρίας τον κύριο Βατλέ και ευελπιστούμε ότι εντός ολίγου θα καταφτάσει και η Επίτροπος Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σας και ελπίζω ότι πραγματικά θα είναι πολύ αξιόλογη μέρα για όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νταϊάννα <clears throat> για αυτή την πολύ εκτενή εισαγωγή και θέλω να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να δώσω το λόγο εις τον κύριο ε, Μελχιόρ ε, ε, Βατλέ που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία με αυτή τη συνάντηση μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναφέρω τις πρόοδους που κάναμε κατά την Βελγική Προεδρία που δεν είναι παρά μόνο ένας σταθμός για να διευκολύνουμε την ζωή των ευρωπαϊκών οικογενειών και ε, σε τομέα του αστικού δικαίου και οικογενειακού δικαίου και εδώ θα τονίσω τα επιτεύγματα της Βελγικής Προεδρίας και σας ευχαριστώ διότι όταν βλέπω το πρόγραμμα που έχετε σήμερα με τον αριθμό των συμμετεχόνων πιστεύω ότι θα έχετε μία μακριά μέρα με πάρα πολλές παρεμβάσεις και νομίζω ότι όλα αυτά τίνουν στο να διευκολύνουν τη ζωή ζωή των Ευρωπαίων από πλευρά αστική. διότι οι Ευρωπαίοι κινούνται όλο και περισσότερο και ευτυχώ, γιατί αυτό επιζητούσαμε ήταν ένα στόχο της Ευρωπαϊκή Ενώσεω και λειτουργεί σωστά άρα ο αριθμός των διεθνών γάμων και των διεθνών σχέσεων ε, καλημέρα σα ε, κυρία Επίτροπε ο αριθμός των διεθνών γάμων αυξάνεται και αυτό είναι θετικό στοιχείο διότι για λόγους επαγγελματικούς, για λόγους ε, πολιτιστικούς, για να μπορέσει κανείς να καλύψει όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν τη δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης, διακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο και περισσότερες διεθνείς ε, καταστάσεις δημιουργούνται, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ανταποκριθούμε από πλευρά αστικού δικαίου και αυτός είναι ο στόχος της σημερινής συνεδριάσεώς μας. Δηλαδή να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί για να τα λύσουμε όσο το δυνατόν πιο διεθνώς διότι όλοι ξεκινήσαμε από την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει όλες αυτές οι διαφορές να μπορούν να επιληθούν. Σήμερα το πρωί λοιπόν μαζί σας θέλω να τονίσω τέσσερα στοιχεία της Βελγικής Προεδρίας και πρέπει να σας πω ότι μπορέσαμε να προχωρήσουμε και να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Καταρχάς την ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά το, την νομοθεσία που εφαρμόζεται σε το διαζύγιο, δηλαδή ε, το οικογενειακό δίκαιο στην Ευρώπη και και για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας όπως προβλέπεται στις συνθήκες και αυτή η πρώτη ενισχυμένη συνεργασία θα λάβει χώρα στο οικογενειακό δίκαιο, τουλάχιστον αυτό εύχομαι, για να καθορίσουμε το τι δίκαιο θα εφαρμόζεται στα διαζύγια. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτή η πρεμιέρα γίνεται κατά τη Βελγική Προεδρία εις το οικογενειακό δίκαιο και στα πλαίσια της ενισχυμένης ε, συνεργασίας για να καταρτήσουμε αυτό το δίκαιο που θα εφαρμόζεται στα διαζύγια θελήσαμε να εξετάσουμε ένα στοιχείο και να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία και να προχωρήσουν για να γνωρίζουν ποιο δίκαιο πρέπει να διέπει το δικαίωμα διαζυγίου να μπορέσουν να το πράξουν. Δηλαδή όλες οι χώρες να ενημερώνονται κατά τρόπον ώστε όλο και περισσότερα κράτη να μπορούν να συμμετάσχουν ε, σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των ε, Ευρωπαίων συνεργατών. θέλαμε να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι νομοθέτης, συνομοθέτης με το Συμβούλιο πρέπει να συμμετάσχει και γι' αυτό θελήσαμε να προχωρήσουμε στο δίκαιο που θα διέπει τα διαζύγια και για συγκεκριμένο λόγο διότι τώρα τα 16 εκατομμύρια ζευγαριών που συνάπτουν γάμο ή ε, την Ευρώπη εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έχουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια ως προς το δίκαιο το οποίο θα εφαρμόζεται στα διαζύγια τους και αυτό τους δίνει μία ασφάλεια. Θέλαμε λοιπόν ε, να ε, τους διευκολύνουμε ως προς την επιλογή τους του δικαιώματος και αν δεν συμφωνήσουν για το δικαίωμα επιλογής του εις νομοθεσίας πρέπει να υπάρχει μηχανισμοί που να καθορίζουν ε, το ε, εφαρμοστέο δίκαιο από τον χώρο διαβίωσης ε, των συζύγων και αυτό δίνει τη δυνατότητα στα άτομα τα οποία χωρίζουν και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουν να πάρουν διαζύγιο με τη μεγάλη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια διότι εάν επιληθεί αυτή η διαμάχη σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο υπάρχει ένα πρόβλημα λιγότερο και μπορεί κανείς να καθησυχάσει την κατάσταση της διαμάχης ε, μέσα στο, στο ε, ζευγάρι για να υπάρξουν και λιγότερα προβλήματα ε, που θα πλήξουν τα παιδιά. Θέλαμε όμως να ασχοληθούμε και με τις κληρονομιές γιατί υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ζουν κάπου αλλά δεν, ε, ε, δεν ε, ε, πεθαίνουν εκεί διότι όπως σας είπα κινούνται στην Ευρώπη και ενδεχομένω έχουν περιουσιακά στοιχεία σε ολόκληρη την ε, ευρωπαϊκή επικράτεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η πραγματική αναγνώριση της ε, αυθεντικής, αυθεντικής περιουσίας για να υπάρχουν λιγότερα θέματα κληρονομικά και να μην είναι αδύνατον να συνεπάρξουν τα διάφορα ε, ε, δίκαια τα οποία δεν συνάδουν υποχρεωτικά πάντοτε στα θέματα κληρονομιάς. Θέλαμε να προχωρήσουμε ε, ακόμη και αν ορισμένα κράτη είχαν δυσκολίες για να προχωρήσουν στο θέμα της κληρονομιάς αλλά το αντάλλαγμα ήταν να μας επιτρέψει επιτρέψουν για να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα να προχωρήσουμε και στο κληρονομικό. Ε, ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι οι απαγωγές των παιδιών διότι η απαγωγή παιδιού όταν ένας από τους ε, δύο γονείς δεν δέχεται ο άλλος να βλέπει τα παιδιά είναι μια τραγική κατάσταση και είναι μια πολύ έντονη κατάσταση γι' αυτό και το παιδί είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο πράγμα το οποίο δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το θέμα επιπλέον ποιες είναι οι λύσεις που πρέπει να επιζητηθούν πώς θα αντεπεξέλθουμε από αυτές τις καταστάσεις κρίσεως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αν προσθέσετε σε αυτό και την, διεθνή διάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο γι' αυτό και σε ε, βέλγικο επίπεδο ε, έχουμε καταρτήσει ένα σύστημα μεσολαβήσεως κατά τρόπον ώστε οι γονείς να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να διαπραγματευτούν, να μιλήσουν μεταξύ τους και να χρησιμοποιήσουμε αυτό το βελγικό σύστημα και στην Ευρώπη για να έχουμε 10 πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα αξιοποιήσουν και θα προκαλέσουν αυτήν την μεσολάβηση όλο και περισσότερο μεταξύ ζευγαριών όταν πρόκειται για διεθνείς καταστάσεις ή για απαγωγές παιδιών. Βέβαια η μεσολάβηση δεν θα λύσει τα πάντα αλλά μπορεί να προλάβει ορισμένα θέματα κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν οι γονείς να δεχθούν το τι μέλη γενέστε. Και ε, στις απαγωγές των παιδιών καταρχήν καταρχήν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των γονιών και ε, ε, το άτομο που ε, είναι εχμάλωτο σε αυτή την κατάσταση είναι το παιδί. Γι' αυτό και χρειάζεται η μεσολάβηση η οποία μπορεί να επιτρέψει να καταλήξουμε σε μία λύση και τα δέκα πιλωτικά προγράμματα τα οποία καταρτήσαμε δείχνουν ότι μέσω της μεσολαβήσεως μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη και στις απαγωγές παιδιών. Και τελευταία τελευταίο θέμα α, όσον αφορά τις, ε, ε, ε, τις διατροφές υπάρχουν πολλά θέματα γλωσσικά, αρχικέ, αρχές υπεύθυνες συνθήκη της Χάγης για την καταβολή της διατροφής και γι' αυτό η Προεδρία του Βελγίου έχει διατυπώσει ορισμένες προτάσεις προς συζήτηση Βλέπετε λοιπόν, είτε πρόκειται για τις απαγωγές, είτε πρόκειται για τα κληρονομικά, είτε πρόκειται για την καταβολή ε, των, της διατροφής, σαν ε, Βελγική Προεδρία προωθήσαμε τα θέματα αυτά ακόμη περισσότερο όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου που θα εφαρμόζεται ε, σε περίπτωση διαδικτύου και σε περίπτωση απαγωγής παιδιών αλλά επαναλαμβάνω ότι ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη πάντοτε διστάζουν να δεχθούν να υπάρξουν άλλες νομοθεσίες που εφαρμόζονται εις το δίκαιο μας διότι ίσως θεωρούμε ότι το άλλο δίκαιο δεν είναι τόσο τέλειο όσο το δικό μας αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι δισταγμοί διότι αυτοί θα είναι εις βάρος της ζωής των ευρωπαϊκών οικογενειών και των ευρωπαίων πολιτών διότι θα υπάρχει υπάρχει επιπλέον μία νομική διαμάχη σε δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις και διαμάχες. Πρέπει να τους διευκολύνουμε, να συνεργαστούμε περισσότερο, να συνάδουν τα αστικά δίκαιά μας και να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για να μπορούν να κινηθούν, να κυκλοφορήσουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλάβουν τις ευθύνες του σωστό αστικό μας δίκαιο και γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και γι' αυτό τα θέματα τα οποία προωθήσαμε κατά την Βελγική Προεδρία είναι στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ότι το ίδιο θα γίνει και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε ε, Υφυπουργέ για τα σχόλιά σας. Καταρχήν θέλω τώρα να χαιρετήσω την κυρία Ρέντινγκ η οποία είναι η Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης και να της δώσω το λόγο ε, ιδίως ευχαριστώντας της που αντιμετώπισε τις καιρικές συνθήκες. Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση που μιλάω ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και βεβαίως πρέπει να σας πω εν παρόδο ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, όλες οι ε, θεσμικές πλευρές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, να υπάρχει δηλαδή στενή συνεργασία ανάμεσα και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εθνικά κοινοβούλια. Τα ζητήματα τα οποία καλούμεθα σε ενωσιακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε είναι παρόμοια και αναφέρονται στους ίδιους ανθρώπους. Έχουμε 12 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή ε, που ε, εφαρμόζουν το δικαίωμά τους να κινηθούν ελεύθερα και να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα και επομένως δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν προβλήματα στις άλλες χώρες. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να αισθάνονται στο σπίτι τους οπουδήποτε και αν πηγαίνουν, οτιδήποτε και αν αποφασίσουν να κάνουν και να ξέρουν ότι έχουν καθήκοντα, υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα. <clears throat> Τι έχει αλλάξει και γιατί κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με την νέα συνθήκη της Λισαβόνας με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Από το 2009 λοιπόν η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με νομικά ε, ζητήματα έφυγε από τα χέρια ε, των ε, Υπουργών των εθνικών χωρών και πλέον μοιράζονται τις αρμοδιότητες αυτές ε, με το Εθνικό Κοινοβούλιο και φυσικά ε, και με την αρρωγή και το, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κάνει κάποια ε, πρόταση και το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν συνομοθέτες σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια αποφασίζουν τελικά επί του πραχθέντος και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι εκεί για να βλέπει εάν οτιδήποτε έχει αποφασιστεί εφαρμόζεται σωστά. για μένα η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και πρέπει να πω ότι κάποια πράγματα ήταν αρκετά εύκολα όταν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Ας πούμε το δικαίωμα των ε, ανθρώπων οι οποίοι συλλαμβάνονται από την αστυνομία και ε, προσαγάγονται ενώπιον της ε, δικαιοσύνης. Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις όσον αφορά ας το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και οι αποφάσεις ελήφθησαν σε χρόνο ρεκόρ και την επόμενη εβδομάδα θα, έχει, θα αποφασιστεί επίσης μια επιστολή ε, <clears throat> κατάλογος δικαιωμάτων. Επίσης η δυνατότητα χρήσης νομικής αρρωγής, η δυνατότητα χρήσης νομικού συμβούλου, ε, δικηγόρου. Αυτά είναι τα ελάχιστα ε, δικαιώματα τα οποία είναι διασφαλισμένα για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη, οπουδήποτε και αν βρίσκεται και αντιμετωπίσει πρόβλημα. Αλλά βεβαίω δεν μα ενδιαφέρει μονάχα να αντιμετωπίσουμε αυτού που βρίσκονται ενώπιον των δικαστηρίων. Ε, θέλουμε να προστατέψουμε και τα θύματα, θύματα ατυχημάτων α πούμε, τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς όταν έχουν ε, υποστεί το ατύχημα αυτό ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη σε μια γειτονική χώρα και όχι στη χώρα στην οποία ζουν. Επομένως μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα συνολικό πακέτο, μια συνολική δέσμη ε, ήπιας νομοθεσίας για την προστασία των θυμάτων. Το ίδιο ε, συμβαίνει και με, την, με τα παιδιά. Θέλουμε μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, γιατί πολύ συχνά τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο εξειδικευμένων προβλημάτων, όταν ας πούμε θα πρέπει να βρεθούν ως μάρτυρες ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα σε μια χώρα που δεν είναι η δική τους. Είμαι θα απολύτως πεπισμένη και αποφασισμένη να εφαρμόσουμε σαν απτή πραγματικότητα τη δυνατότητα ε, κυκλοφορίας των, ε, και, και ε, κυκλοφορία συγγνώμη, των πολιτών. Είχαμε προκαιρού μια κοινή συνέντευξη τύπου ο κύριος Μισελ Μπαρνιέ, Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και υποφαινομένη ως υπεύθυνη για τους πολίτες και την, το νομικό πλαίσιο. Εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν να πούμε πώς θέλουμε να εμφυσίσουμε νέα ζωή στην ενιαία εσωτερική αγορά, όχι όμως μονάχα από οικονομική άποψη. Οι πολίτες είναι το ίδιο σημαντική, αν όχι περισσότερο, από την οικονομία. Επομένως μας ενδιαφέρουν η οικονομία, αλλά και οι πολίτες γιατί είναι οι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος και αυτό ακριβώς προσπαθεί να καταδείξει και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, ήδη ε, ο κύριος Βουατλέ μίλησε για το κληρονομικό δίκαιο ε, και βεβαίως υπάρχουν ε, ακόμα κι άλλα προβλήματα 450.000 περίπου περιπτώσεις κληρονομικού, διασυνοριακού κληρονομικού δικαίου αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο και επομένως βεβαίως θέλουμε εναρμόνιση του εφαρμοστέου δικαίου ε, χρησιμοποιώντας την, τον συνήθι τόπο διαβίωσης ε, σαν βάση και βεβαίω θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μονάχα ένα δικαστήριο θα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του κληρονομικού ε, δικαίου και ότι θα διέπονται όλοι από ένα ενιαίο δίκαιο. Και επίσης η απόφαση δικαστηρίου ενός που έχει ληφθεί σε μία χώρα μέλη θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό σαν επίσημο έγγραφο από ένα άλλο δικαστήριο και επομένως να μην χρειαστεί ο ενδιαφερόμενος να περάσει μέσα από νέες διαδικασίες σε κάθε μεμονωμένη καινούργια χώρα μέλος έτσι ώστε να ξαναπάρει αυτό το ε, ε, πιστοποιητικό. Ε, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως επίσης το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Κληρονομίας είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ε, γιατί θα διασφαλίσει ε, περισσότερο τα κληρονομικά δικαιώματα δεν τα δικαιώματα των κληρονόμων, αλλά θα διευκολύνει ε, και την άσκηση δικαιωμάτων των ε, πολιτών χρησιμοποιώντας ένα και μόνο έγγραφο σε όλες τις χώρες μέλη και θα διευκολύνει φυσικά και γραφειοκρατικά και τις διάφορες υπηρεσίες. Η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προσπαθούν να δουν τις λεπτομέρειες της πρότασης αυτής και είναι αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται φυσικά πολύ στενά με τους ε, συνομοθέτες έτσι ώστε να ε, προκύψει μια κατάσταση νομικής βεβαιότητας και νομικής ασφάλειας ε, την οποία οπωσδήποτε χρειάζονται οι ε, πολίτες. Μέχρι τώρα οι επαφές που είχαμε με τον κόσμο και η μελέτη αντικτύπου έχουν δείξει ότι αναμένουν οι πολίτες με μεγάλη προσδοκία τις αποφάσεις και είμαι βεβαία ότι θα, μπορέσουμε να βρούμε τελικά μια συμφωνία η οποία θα είναι αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό είναι ένα μονάχα από τα στοιχεία τα οποία αφορούν τους ε, πολίτες, ε, διότι τελικά εκείνοι θα επωφεληθούν ε, περισσότερο από τα δικαιώματα τα οποία θα συνδέονται με την κινητικότητά τους και το δικαίωμα κινητικότητας που έχουν. Όσον αφορά όμως και τα ε, ζευγάρια, τα παντρεμένα ή μη, βεβαίως θέλουμε πρόθεση του γαμικού δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα διεθνή ζευγάρια να γνωρίζουν ποιος είναι ο νόμος, ποιο είναι το δίκαιο το οποίο ε, θα εφαρμοστεί στη δική τους περίπτωση, ποιος είναι ο νόμος που θα διέπει ε, την περιουσία τους. Αναγνώριση λοιπόν των ε, ε, περιουσιακών τους στοιχείων και των περιουσιακών τους δικαιωμάτων ε, όσον αφορά, την, όσον αφορά όλες τις χώρες, δηλαδή να αναγνωρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα δικαιώματά τους σε όλες τις χώρες. και επομένως ε, περιμένουμε επίσης ε, και με πολύ μεγάλη ε, προσδοκία και τον νέο κανονισμό όσον αφορά το διαζύγιο. Να σας εξηγήσω και κάτι. Ο κανονισμός για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο είναι η πρώτη απόφαση η οποία λαμβάνεται επί τη βάση ενισχυμένης συνεργασίας. Σαν Λουξεμβούργια δεν είμαι πολύ υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας. Εγώ ε, νομίζω ότι είναι καλύτερα ε, να προχωρούν και 27 χώρες μαζί και όχι μονάχα μία ομάδα και μου χρειάστηκε πολύς χρόνος πριν αποφασίσω ότι παρόλα αυτά έπρεπε να προχωρήσω προς την ε, κατάσταση αυτή. Είναι ε, μια, ε, πραγματικά είναι μια πρώτη φορά ε, που προτείνεται μια τέτοια διέξοδος έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αδιέξοδα και εμπλοκές όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόκειται για μια ανοιχτή, ενισχυμένη πλειοψηφία, επομένως όλες οι χώρες, εάν επιθυμούν, μπορούν να μπουν στη διαδικασία αυτή, αλλά έπρεπε να γίνει μια επιλογή ανάμεσα στο να υπάρχει μια λύση για τις, τους περισσότερους πολίτες μέσω αυτής της ενισχυμένης ε, ε, συνεργασίας να καλύπτονται δηλαδή τουλάχιστον κάποιοι πολίτες ή από την άλλη πλευρά ε, η επιλογή να μην υπάρχει καμία λύση για κανέναν πολίτη και επομένως να συνεχίσουν να υφίστανται τα προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίων διασυνοριακών. Σε αυτή την περίπτωση αποφασίσαμε ότι η ενισχυμένη πλειοψηφία θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερη επιλογή. Ε, και μια τέτοια διαδικασία θέλησαμε να ακολουθήσουμε ε, και για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας γιατί ακριβώς μπορεί να δώσει διέξοδο σε μια κατάσταση εμπλοκής. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εγγράφων αποτελεί βεβαίως προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία. Ας πούμε, πιστοποιητικό γεννήσεως χρειάζεται για να γραφτεί ένα παιδί στο σχολείο ή για να ε, ε, ε, μπορεί κανείς να έχει, να έχει κάποια βοήθεια από το κράτος για τα παιδιά που έχει ή ε, για την κοινωνική του ασφάλιση ή για να αναγνωριστεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή όμως έγγραφα τα οποία αναγνωρίζονται μονάχα ε, στον τόπο έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού. Επομένως ε, θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση το Δεκέμβριο ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά τα οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικά. Θα λάβουμε φυσικότατα υπόψη και θα αποτελέσει σημαντική συμβολή σημερινή σας συζήτηση και θα προτείνομαι λοιπόν δύο νομικού περιεχομένου προτάσεις όσον ε, αφορά ε, την αναγνώριση δημοσίων εγγράφων και όσον αφορά την αναγνώριση ε, του καθεστώτος υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βρίσκονται ε, μέσα στο, στο, στο κέντρο, στο επίκεντρο της διαμάχης των γονιών τους, οι οποίοι ε, προέρχονται από διαφορετικές χώρες ε, και πρέπει να πούμε ότι στο άρθρο 14 του Χάρτας Θεμελιδών Δικαιωμάτων γίνεται συγκεκριμένη και ρητή αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών και επομένως θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις διαφορές αυτές να επιληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπέρ των παιδιών. Η απόφαση, και η εφαρμογή ε, των αποφάσεων σχετικά με, ε, ε, σχετικά με την γονική ημέρημνα θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί. Φυσικά υπάρχει η υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά την αναγνώριση των γονικών δικαιωμάτων αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά προσκόμματα όσον αφορά την την υποχρέωση εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών σε άλλη χώρα από αυτήν στην οποία έχουν εκδοθεί. Ε, επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε και τις περιπτώσεις απαγωγής παιδιών και διασυνοριακής απαγωγής παιδιών. Αυτά που ανέφερα κυρίες και κύριοι είναι μονάχα κάποια από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν αλλά βλέπετε όλοι ότι έχουμε επιταχύνει τη διαδικασία. Έχουμε περάσει στην επόμενη ταχύτητα η χρήση της εσωτερικής αγοράς ε, σαν ε, χώρου ελεύθερης επιλογής των ε, πολιτών μας. Δεν θα πρέπει να παραμείνει μονάχα δικαίωμα στα χαρτιά. Θα πρέπει να γίνει δικαίωμα στην πράξη. Θα πρέπει να ξεπεραστούν όλα τα προσκόμματα τα οποία, έχουμε, ε, τα οποία αντιμετωπίζομαι ε, μέχρι τώρα. Ε, η Κομισιόν θα προτείνει λοιπόν και στο μέλλον έτσι ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συναποφασίσουν υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να αποφασίσουν λέγω μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε αποφάσεις και ελπίζομαι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό το, το εννιάμινο διάστημα είναι εξαιρετικά σύντομο για, τον, ε, για το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα έτσι ώστε τα 12 εκατομμύρια άνθρωποι στους οποίους αναφερόμαστε να λύσουν τα προβλήματά τους και να έχουν ασφάλεια δικαίου. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τα σχόλιά σας. Τώρα ξεκινάει η πρώτη συνεδρίαση εργασίας και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Ταντέους Βίρκα ο οποίος είναι ο συντονιστής της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Συντονιστής. Έχεις το λόγο Ταντέους. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να απευθύνω θερμό καλωσόρισμα προς όλους τους συμμετέχοντες και να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή συνάντηση σε αυτή τη Σύνοδο Εργασίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους βουλευτές και γερουσιαστές από τα Εθνικά Κοινοβουλευτικά Σώματα και τους Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα όλος ιδιαίτερος και εγκάρδια να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους ε, πανελίστες μας, ε, τους προσκεκλημένους που θα μας διαφωτίσουν με την πλούσια πείρα και γνώση τους, γιατί το φάσμα είναι τεράστιο και εξαιρετικά ευρύ, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ευαίσθητο και πολύ λεπτό, γιατί άπτεται περίπλοκα θέματα του οικογενειακού δικαίου. Θα ήθελα ταυτόχρονα να καλωσορίσω και τον Μάρκο Ντιές Δεσέρα, τον κύριο Γερουσιαστή που ε, είναι αρμόδιος για θέματα νομικά στην ε, Ισπανική Γερουσία και θα είναι ο πρόεδρός μας ε, σε αυτό το πάνελ και μάλιστα κατά το πέρας της συζήτησης θα μας κάνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί βουλευτέ, γερουσιαστέ και ευρωβουλευτέ, ότι έχετε λάβει διάφορα όργανα και όποιος θέλει να λάβει το λόγο μπορεί να το δηλώσει στη διάρκεια των ομιλιών που θα ακούσουμε ώστε να διοργανώσουμε και τη διεξαγωγή της συζήτησης. Αυτό είναι απαραίτητο διαδικαστικό θέμα γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία 20 καθυστέρηση οπότε θα ήθελα να αφιερώσουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στη συζήτηση για να ακούσουμε τις απόψεις των εθνικών βουλευτών να μας εκφέρουν τη θέση τους, να υποβάλουν τις απορίες τους, ώστε να είναι όσο πιο επικοδομητική και καρποφόρα γίνεται η σημερινή συνάντηση. Ως μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθημερινά αντιμετωπίζω επίμαχα θέματα οικογενειακού δικαίου. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσω και τις ε, παρεμβάσεις των εμπειρογνωμόνων μας γιατί όντως είναι ένα θέμα περίπλοκο και συγκινησιακά φορτισμένο το θέμα του οικογενειακού δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να, να ζητήσω θερμά και από τους εμπειρογνώμονές μας να τηρήσουν το χρόνο αγόρευσης. Θα ήθελα ο καθένας να τηρήσει αυστηρά και βλεβικά το δεκάλεπτο παρακαλώ για να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα ενδιαφέροντα για μας θέματα. Ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι η Κατερίνα Μπελβέλκη, καθηγητής ε, Δημοσίου Ιδιωτικού Δικαίου ε, και Οικογενειακού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Η κυρία Βέλκη θα μας ε, υποβάλει το θέμα της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας για θέματα διασυνοριακών γάμων, την πρόταση δηλαδή Ρώμη 3, που αναφέρθηκε και πριν από λίγο. Το λόγο έχει η καθηγήτρια από την Ουτρέχτη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της πρόταση για το Συμβούλιο Συμβουλίου και Επιτροπή για την ενισχυμένη συνεργασία, διευρυμένη συνεργασία σε εφαρμοστέο δίκαιο σε θέματα διαζυγίου και χωρισμού νομικού. Η πρόταση με τον τίτλο Ρώμη 3 περιλαμβάνει ενιαίες διατάξεις ε, για, το για διασυνοριακά θέματα σε περίπτωση ο μελλοντικό ε, κανονισμό ε, Ρώμη 3 θα τεθεί σε ισχύ μόνο για 14 χώρε μέλη. Όπω ακούσαμε, για πρώτη φορά σε θέματα συνεργασία αστικού δικαίου εφαρμόζεται σε διαδικασία διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, 13 χώρε μέλη δεν θα συμμετέχουν, δεν θα εγκρίνουν τον κανονισμό Ρώμη 3 και θα εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους ε, εθνικούς κανόνες ε, για τη σύγκρουση δικαίου, που είναι διαφορετική από τους κανόνες του Ρώμη 3. Παρόλο που το 2008 είχαμε συμφωνία για την προηγούμενη πρόταση Ρώμη 2, η... για την πρόταση Ρώμη 3 δεν υπήρξε πλήρη συμφωνία. Εγώ δεν θα σας αναλύσω αυτή τη διαδικασία του κανονισμού Ρώμη 3, αλλά θα θέσω κάποια ερωτηματικά για το περιεχόμενο της πρότασης Ρώμη 3. Καταρχήν είναι σημαντικό ότι οι σύζυγοι ορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο. Το θέμα είναι πότε θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβούν στην επιλογή τους. Σύμφωνα με την πρόταση Ρώμη 3 δεν υπάρχουν περιορισμοί στο χρόνο επιλογής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας, ενός γαμικού συμβολέου που συνήθει στην αρχή του γάμου και ενός συμβολέου ε, διαζυγίου γιατί το πρώτο συμβόλαιο είναι δεσμευτικό για το εγγύς και απότερο μέλλον και η σύνδεση μεταξύ του νόμου του δικαίου που επιλέχθηκε την στιγμή της συμφωνίας ίσως να μην υπάρχει στη στιγμή του διαζυγίου, του χωρισμού. Οπότε οι σύζυγοι θα πρέπει να κάνουν πιο ε, εμπεριστατωμένες και σωστές ε, αναλύσεις τη στιγμή που αποφασίζουν να λύσουν τη γαμική του σχέση, όχι τη στιγμή της σύναψης του γάμου, γιατί η στιγμή της διάλυσης του γάμου μπορεί να λάβει χρόνια, πολλά χρόνια μετά τη σύναψη του γάμου. Οπότε είναι λογικό και πιο ε, επίκαιρο να αποφασίζουν τη στιγμή της ε, λύσης του γάμου. Βέβαια, το γεγονός της υπογραφής και ημερομηνία από τους δύο σύζυγους δεν είναι σίγουρο ότι εξασφαλίζει τη γνώση των σύζυγων. Γιατί δεν ε, είναι υποχρεωτική η νομική συμβουλή. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχουν νομικές ε, πληροφορίες ε, που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, είναι μερικές φορές δυσνόητες, οπότε είναι σκόπιμο να προσφύγουν σε νομική συμβουλή Γι' αυτό ισχύει και για τις πληροφορίες που δίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για τη Δικαστική Συνεργασία. Επίσης δεν αναφέρεται γιατί η πρόταση Ρώμη 3 μιλάει για το τελευταίο ρόλο διαμονής, της κοινή διαμονής. Αυτό βέβαια υπόκειται στον όρο ότι ένας από τους συζύγους εξακολουθεί να παραμένει εκεί και υπό κάποιες συνθήκες η κοινή διαμονή δεν θα πρέπει να έχει σταματήσει ένα χρόνο πριν την απόφαση του δικαστηρίου. Βέβαια, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων. Και αν δεν δοθεί από χρόνο λόγος για το γιατί αυτός ο περίπλοκος συνδετικός κρίκος χρησιμοποιείται για, την, για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, θα πρέπει η σχετική διάταξη να διαγραφεί. Γιατί έτσι οι διατάξεις εφαρμοστέου δικαίου, το άρθρο 3 και 4 της, του κανονισμού Ρώμη 3, θα είναι πιο εύκολες στην πράξη ένα από τα βασικά επιχειρήματα ορισμένων κρατών μελών για να μην ε, ε, εμπλακούν στην ε, διευρυμένη συνεργασία είναι ότι ίσω η σύγκρουση δικαίου οδηγήσει στην εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου. Ο κανονισμό όμω Ρώμη δέχεται αυτή την έκβαση, αλλά προβλέπει κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε. Για παράδειγμα, το διαδικαστήριο ενό από τα κράτη-μέλη δεν θα εφαρμόσει ε, διατάξει με διακριτική μεταχείριση. Επίσης, οι θεμελιώδες ε, αρχές και δικαιώματα θα πρέπει να παραβιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης έχει την υποχρέωση να προσδιορίσει από την αρχή ποια ε, δίκαια διαζυγίου του παγκόσμιου συστήματος δια ή καταστρατηγούν την αρχή ίσης πρόσβασης ε, στο διαζύγιο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τρεις διατάξεις της Ρώμης 3 λαμβάνουν υπόψη ότι ούτε διαζύγιο ούτε λύση ε, γάμου μετά, τη νομική, μετά το νομικό χωρισμό μπορεί να γίνει στη Μάλτα. Και τα διαζύγια των υπόλοιπων χωρών πριν της Μάλτας μπορούν να εφαρμόσουν το, το, τη διάταξη 3 αλλά τα μαλτέζικα δικαστήρια δεν μπορούν να υποχρεωθούν να εκδώσουν διαζύγιο, ακόμη και αν άλλο αλλοδαπό δίκαιο για το διαζύγιο στην περίπτωση αυτή είναι εφαρμοστέο. Είναι πραγματικά λυπηρό που τα άλλα συμβαλόμενα μέρη της ε, διευρυμένης συνεργασίας δεν ε, ε, απέρριψαν την συμπερίληψη μιας τέτοια διάταξης σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί υιοθετούν ένα τελείως εθνικό πρίσμα και οι διατάξεις για τη Μάλτα είναι ένα πιστοδρομικό βήμα ε, που πλήττει τις διατάξεις για το διαζύγιο στην Ευρώπη και δίνουν πολύ ασφαλμένο μήνυμα. Η γενική μου εκτίμηση για την πρόταση ρομετρή είναι αρνητική. Και παρά την δυνατότητα που έχουν οι σύζυγοι να καθορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο, οι διατάξεις είναι γενικώ περίπλοκες και δυσεφάρμοστες. Η δομή της πρότασης δεν είναι πιστική, θα μπορούσε κάλλιστα να βελτιωθεί. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι οι σημερινές επιλογές είναι πολύ σχετικές για το μέλλον. Δεν θα πρέπει να δεσμευτούμε από τώρα για το μέλλον, γιατί στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερες ε, ε, ιδιωτικές ρυθμίσεις σε διασυνοριακά θέματα. Οπότε για θέματα ε, Συνοχή, θα λαμβάνεται υπόψη η Ρώμη 3, θα δίνει δηλαδή τη βασική κατεύθυνση. Εγώ θα προτιμούσα να υιοθετήσουμε το Lex Fore ε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαφορετική επιλογή των ε, συζύγων. Βέβαια το επιχείρημα ότι το, η εφαρμογή του Lex 4 θα οδηγήσει σε τουρισμό διαζυγίου, γιατί σε ορισμένες χώρες είναι πιο εύκολη η έκδοση διαζυγίου από ό,τι σε άλλες, δεν είναι... Ε, βάσιμο επιχείρημα, γιατί η Ρώμη 3 δεν είναι απομονωμένη πρόταση. Η Βρυξέλλες 2α που αφορά τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου λαμβάνεται επίση υπόψη. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει αποδειχθεί ότι με βάση το καθεστώς των Βρυξελών 2α οι, σύζυγοι χρησιμοποιούν διάφορες δικαιοδοσίες προκειμένου να διευκολυνθούν στην έκδοση διαζυγίου σε χώρες που δεν έχουν, με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση. Η Ρώμη 3 λοιπόν δεν θα επιλύσει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Για αυτούς και για άλλους λόγους που παραθέτω στο έγγραφό μου θα σας πρότεινα να μην εγκρίνετε την πρόταση Ρώμη 3. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Τα θέματα τα σχετικά με τον κανονισμό Ρώμη 3 είναι εξαιρετικά περίπλοκα και όντως θα είναι περιορισμένη η εφαρμογή του κανονισμού αυτού Ρώμη 3. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι είναι αξιόλογος αυτός ο κανονισμός και έχει μια προστιθέμενη αξία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην διαδικασία αυτή έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά είμαστε ευγνώμονες προς τη Βελική Προεδρία που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ε, φαίνεται και στη συνεδριάση του Κορεπέρ. Θα έχουμε τη δυνατότητα πάντως να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συζήτηση για το θέμα αυτό και να δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο εμπειρογνώμονά μας, στον κύριο Σχεφ Βαν Έρπ, τον καθηγητή αστικού και ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου στο, Πανεπιστήμιο, στο Ινστιτούτο Ιδιωτικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Μάστριχτ και επίσης ε, δικαστή στο εφετείο του Χόρκεμπος ο κύριος Βανέρκ θα μας μιλήσει για θέματα περιουσιακών σχέσεων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι να κάνω κάποιες προκαταρτικές ε, ε, παρατηρήσεις. Όταν μιλάμε για διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, βεβαίως αναφερόμαστε και σε διασυνδέσεις με, το, ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και με δικαιώματα όπως η ελευθερία, και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε δηλαδή το ιδιωτικό δίκαιο από άλλα ε, ε, δικαιώματα. Ας πούμε, το δίκαιο το οποίο διέπει το, το γάμο δεν μπορεί να χωριστεί από το κληρονομικό δίκαιο. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω όμως την προσοχή μου στην ε, σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό δίκαιο και το ουσιαστικό δίκαιο. Όχι γιατί πρόκειται για αντιφατικά συστήματα, αλλά γιατί θα πρέπει να ρωτηθούμε αυτή τη στιγμή ε, πώς μπορούμε να συντονίσουμε ε, διαφορετικά δίκαια, ε, πώς μπορούμε να συντονίσουμε και να διευκολύνουμε επομένως τη ζωή ανθρώπων που εργάζονται συνοριακά ή παντρεύονται διασυνοριακά ο τρόπος που επιλέγουν οι άνθρωποι να συζήσουν ε, είναι περίπλοκος. Πρώτα απ' όλα μπορούν να συζήσουν χωρίς ε, να ρυθμίσουν τίποτα, δηλαδή χωρίς να πατρευτούν, αλλά χωρίς ε, και να συνάψουν οποιοδήποτε συμφωνία συμβίωσης. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόζεται το ιδιωτικό δίκαιο. Δηλαδή, να ε, αν μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία. Εάν κάποιος λοιπόν από τη Γερμανία αρχίσει να ζει ε, με κάποιον από το Βέλγιο, τότε θα πρέπει το αλλάζουν στο Βέλγιο, τότε, θα, τότε ε, τα ε, στοιχεία τα οποία βρίσκονται, περισσότερα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο Βέλγιο θα, θα διέπονται από το βελγικό νόμο, τα υπόλοιπα από τον γερμανικό, γιατί ο ένας από τους δύο είναι γερμανός. Επομένως θα πρέπει να αποφασίσει, αποφασίσουν οι ίδιοι ποιοι, ποιος θα είναι ο εφαρμοστέος νόμος, ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Ε, και έχουν τη δυνατότητα για ένα περίεργο λόγο να επιλέξουν σαν εφαρμοστέο δίκαιο το γαλλικό δίκαιο. Επομένως θα πρέπει να απλουστεύσουμε λίγο τις διαδικασίες αυτές. Ε, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν λίγο εάν ε, συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. Τότε επιλέγουν και ένα καθεστώς και επομένως ε, εφαρμόζεται το δίκαιο ε, της ε, χώρας όπου έχει συναυθεί ή έχει δηλωθεί αυτή η συμφωνία συμβίωσης υπάρχουν χώρες οι οποίες δέχονται και ε, ε, γάμους μεταξύ ομοφύλων ε, και επομένως σε αυτή την περίπτωση πάλι διέπονται από το δίκαιο στην χώρα, της χώρας στην οποία έχει συναυθεί ο γάμος. Αυτό που θα ήθελα να πω τη στιγμή είναι ότι εάν γίνει κάτι, οτιδήποτε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή εναρμόνιση, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ε, δουν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες το τι έχουν κάνει άλλοι διεθνείς οργανισμοί ε, ή Ινστιτούτα. Γιατί θα ήταν κρίμα να μην ληφθεί υπόψη καθόλου το τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Επομένως, μπορώ να συστήσω τα εξής. Πρώτον, η κινητικότητα των ατόμων δεν είναι μόνο ε, σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής αγοράς αλλά και μέσω έκφρασης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να ληφθούν οι ε, υπόψη ε, το εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά την σύναψη γάμου ή άλλης βεβαιωμένης σχέσης και θα πρέπει οπωσδήποτε να διέπεται από τον από το ιδιωτικό δίκαιο αλλά με τρόπο που να δίνεται στα άτομα ικανοποιητικός βαθμός ελευθερίας και κάλυψης των δικαιωμάτων τους. Οι καταγραμμένες ε, συμβιώσεις θεωρητικώς είναι ε, ε, νόμιμες σχέσεις καταγραμμένες σε μία χώρα. Παρόλα αυτά νομικές έρευνες καταδεικνύουν ότι ε, ενδεχομένως εφαρμόζεται το, το λέγιο εξ πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτού του είδους οι σχέσεις να είναι απολύτως αυτόνομες και επομένως να εφαρμόζεται πλήρως το δίκαιο το οποίο διέπει όλους τους ε, ε, υπόλοιπους εγκατεστημένους ε, στη χώρα αυτή και στην περίπτωση των καταγεγραμμένων συμβιώσεων. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε οποιαδήποτε μορφή ε, γάμου. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, να αναλυθούν ε, περαιτέρω κυρίως δε να ληφθούν υπόψη τα περιουσιακά δικαιώματα, το, τα οικονομικά δικαιώματα και όχι μονάχα όπως αυτά αναφέρονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και όπως έχουν μελετηθεί και από άλλα συστήματα. οι περιουσιακές επιπτώσεις της λύσεως μιας καταγεγραμμένης σχέσης ή ενός γάμου ε, θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη. Δεν καταλαβαίνω, ε, δεν υπάρχει εμφανής λόγος γιατί πρέπει να υπάρχει διαφορετικό δίκαιο για την λύση ενός, ενός γάμου ή μιας καταγεγραμμένης επίσημης ένωσης. Ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να πει ότι για περίπτωση λύσεως μόνιμης σχέσης ή ε, γάμου θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη λέγω η πρόταση της Γερμανίας και της Γαλλίας να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ε, λύσης ε, των ε, σχέσεων. Αλλά μπορεί κανείς να διαλέξει, να επιλέξει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο άσχετα από τα πρότυπα τα οποία διέπουν τις μεμονωμένες χώρες ή ε, θα πρέπει να πούμε ότι by default θα εφαρμόζεται ε, το δίκαιο μίας χώρας, την οποία θα επιλέξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε πολλές περιπτώσεις ε, ο ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό δίκαιο ίσως μπορεί να πηγαίνει πιο μακριά. Αλλά παρόλα αυτά ε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εφαρμοστέου δικαίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα διαρκή και συνεχόμενα προβλήματα τα οποία ε, αντιμετωπίζει το αστικό δίκαιο όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση στοιχείων. Μπορεί κανείς να πει ότι ε, η ευρωπαϊκή ε, νόμη αναγνώρισης των ε, περιουσιακών δικαιωμάτων, των κληρονομικών δικαιωμάτων είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιοδήποτε οικονομικές συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί είναι σημαντικός και ο ρυθμός των καταγεγραμμένων ε, επίσημων σχέσεων συμβίωσης. Και εκεί υπάρχει θέμα περιουσιακών σχέσεων, ε, κληρονομικών σχέσεων και σίγουρα μια καλύτερη συνεργασία θα ήταν πολύ θεωρητικό στοιχείο. Αναφερθήκατε στην γαλλογερμανική πρόταση πάνω στην ώρα γιατί αυτό είναι το θέμα της επόμενης παρουσίασης της κυρίας Εύα Μπέικερ που είναι ε, δικηγόρος από το δικηγορικό γραφείο Jugendburth and Becker του Βερολίνου που θα μας παρουσιάσει πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα για ορισμένες πτυχές ε, περιουσιακών γαμικών σχέσεων όπως αναφέρονται στην προαιρετικη γαλλογερμανική πρόταση. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Θέλω να σας αναφέρω κάτι πολύ επικοδομητικό για την Ευρώπη, δηλαδή τη συμφωνία για την, ε, τον τρόπο της ε, κατανομής της οικογενειακής περιουσίας, διότι ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε μία αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των εθνικών δικαίων και γι' αυτό δεν αναφερώ Είμαστε εις το το δίκαιο αλλά εις την συνεργασία της Γαλλίας και της Γερμανίας ή στον τομέα ε, ε, της κατανομής της περιουσίας ε, και έχει επιλεγεί η τον τομεα της νομοθεσία διότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα πραγματικότητα τώρα είναι μένα μία πρόοδος για την Ευρώπη αλλά αποδεικνύει ότι υπάρχει ε, σημαντική και επίγουσα ανάγκη να επιλύσουμε το θέμα των οικογενειακών ε, σχέσεων. Αν αυτό δεν ε, έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρόλο που υπάρχουν και στη γαλλική και στη γερμανική νομοθεσία δυνατότητες οι οποίες λειτουργούν σωστά και ρυθμίσεις χωρίς όμως να καλύπτουν το θέμα διότι ε, δεν έχουν ε, ε, δεν αναφέρονται στο εμπράγματο δίκαιο και υπάρχει και μία διασύνδεση με το εμπράγματο δίκαιο, με το κληρονομικό δίκαιο και τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Έπρεπε λοιπόν λοιπόν να ευρεθεί μία λύση η οποία να εξασφαλίσει τα εξής. Καταρχήν ότι θα μπορούσε η νέα κατάσταση να λάβει υπόψη και τα δύο δίκαια... και να ε, ε, ε, μην άπτεται ακριβώς του εκάστοτε εθνικού δικαίου χωρίς να μειώνει τα δικαιώματα των δύο δίκων. Επίσης έπρεπε να βρεθεί καλύτερη λύση για το οικογενειακό σπίτι που ήταν το πιο σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο και να βρεθεί μια σωστή ρύθμιση από την Επιτροπή που αναφέρθηκε και ανέλαβε την επεξεργασία του ρυθμίσεως αυτού του θέματος ε, έγινε, ε, έγινε ε, μία απογραφή των διαφόρων δικαιωμάτων κατά τρόπον ώστε να μπορούν και τα δύο μέρη να έχουν τα ίδια δικαιώματα και αυτό σημαίνει ότι στην αρχή και στο τέλος της σχέσεως θα πρέπει να υπάρχει μία απογραφή κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία αποζημίωση αντίστοιχη κατά την το διαζύγιο. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ μόνο σε δύο-τρία θέματα ε, για να καταλάβετε τι δυσκολίες αντιμετώπισε η Επιτροπή για να επιλύσει αυτές τις περιουσιακές διαφορές. Καταρχήν υπάρχει δυνατότητα να ε, ρυθμιστεί η οικογενειακή κατοικία από κοινού και υπάρχουν μέτρα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ την γερμανική νομοθεσία αλλά θεωρήσαμε ότι το πιο ουσιαστικό θέμα στις ρυθμίσεις αυτές ήταν ε, το οικογενειακό σπίτι. Ε, μία άλλη ιδιομορφία ήταν στην περίπτωση των δωρεών και σύμφωνα με το άρθρο 8 και 10 της γερμανικής νομοθεσίας προβλέπεται ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι δωρές οι οποίες έχουν γίνει από τους δύο συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου και ε, ε, θα πρέπει ε, να ληφθούν υπόψη δύο χρονικά σημεία τα οποία, ε, να, επί των οποίων να μπορέσει κανείς να καταγράψει την οικογενειακή περιουσία. Βλέπουμε ότι θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τις ανατιμήσεις της αξίας της ε, οικογενείας και ε, να μπορέσει κανείς να καθορίσει επακριβώς την αξία της οικογενειακής περιουσίας στην αρχή και στο τέλος του γάμου κατά τρόπον ώστε ε, να συνυπολογιστούν τα αγαθά και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία η οικογένεια έχει κατά τη στιγμή του χωρισμού και να αφαιρεθούν από αυτά τα ε, κοινά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπήρχαν κατά την έναρξη της έγγαμης σχέσεως και ε, βεβαίως ε, υπάρχουν στα θέματα αυτά ανατιμήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα χωρίς παρέμβαση των συζύγων και πρέπει να βρεθεί ε, μια συμβιβαστική λύση όπως άλλωστε και ένας τρόπος της ε, ε, της, ε, του υπολογισμού της την αριθμικής αναπροσαρμογής και η ρύθμιση αυτή αναφέρεται εις το άρθρο 9 της νομοθεσίας και αναφέρεται τις αλλαγές των τιμών στα διάφορα κράτη-μέλη. Προσπάθησε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να εξετάσει αν σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτή η τιμαριθμική αναπροσαρμογή και εκεί αντιμετώπισε προβλήματα διότι βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει ένα στοιχείο κοινή περιουσίας κατά τις διαδικασίες αυτές και θα έπρεπε να βρεθεί μία εναρμόνιση του εμπράγματου δικαίου διότι ε, τα διαζύγια έχουν πολύ περισσότερο συγκινησιακού παράγοντες παρά ε, μία ε, θέληση εξέβρεσης συμβιβαστικής λύσης. Το πρόβλημα όμως είναι αρκετά σοβαρό και έπρεπε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι εθνικές παραδόσεις γι' αυτό και στις γερμανογαλλικές σχέσεις στον τομέα αυτό ε, βρέθη μία ρύθμιση η οποία είναι είναι και πρακτική ε, και συμφέρουσα ε, και ε, να μπορεί να μετατεθεί και σε άλλες νομοθεσίες πέραν της γαλλικής και της γερμανικής διότι ενδέχεται και άλλα κράτη να ενδιαφερθούν για αυτές τις ρυθμίσεις και έτσι αποφασίσαμε να προβλέπεται στη ρύθμιση συμμετοχή και περαιτέρω κρατών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η συμφωνία για τη ρύθμιση των περιουσιακών στοιχείων είναι διαθέσιμη για όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω να καταφύγει κανείς και πάλι εφόσον συμφωνήσει σε ένα εθνικό δίκαιο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα είναι σκόπιμο η εργασία αυτή να συνεχιστεί προς περαιτέρω εναρμόνιση και να προβλέπεται μια εξασφάλιση των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των εταίρων στην οικογένεια και ε, η γρήγορη λύση. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπέκερ, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι οι εμπειρίες που συλλέξαμε από τη διμερή συνεργασία μπορούν ε, να μεταφερθούν ε, και σε ευρύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις και να αξιοποιηθούν. Χαίρομαι που υπάρχει ήδη τέτοια συνεννόηση και ελπίζω να είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες μέλη αυτή η συνεννόηση, γιατί μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε τη δική σας ερμηνεία από αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Θα ήθελα να κάνω μία τεχνική παρατήρηση για όλους τους συμμετέχοντες. Δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχύουν ιδιαίτερες διατάξεις για την Ολομέλεια. Δεν μπορεί κανείς να φέρει ποτό οτιδήποτε υγρό στην, ε, στην αίθουσα της Ολομέλειας απαγορεύεται, αλλά ακριβώς πίσω από την αίθουσα υπάρχει το γνωστό καφενείο Mickey Mouse, μπορείτε να πιείτε ό,τι θέλετε, καφέ, χυμούς, αλλά παρακαλώ μην φέρετε οτιδήποτε υγρό, ποτό μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, δυστυχώς απαγορεύεται. Εν πάση περιπτώσει μια πρακτική πληροφορία ήταν αυτή και συνεχίζουμε την ακρόασή μας με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα που περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη και τη αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ομοφιλόφιλων γάμων ή θέματα συμφωνιών συμβίωσης μεταξύ είτε ομοφιλόφιλων ζευγαριών είτε ζευγαριών διαφορετικού φύλου. Θα έχουμε δύο εμπειρογνώμονε εδώ. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπεατρί Γκουτ, που είναι πρόεδρο τη Επιτροπή Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο ε, της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και αυτό το λεπτό ζήτημα να σας δώσω τρία μηνύματα. Καταρχήν, μία επισκόπηση που δείχνει μία αταξία, αρκετή αταξία, για να μην πω πολύ σημαντική σε θέματα νομικά και μια βεβαιότητα νομική είναι το δεύτερο μήνυμα, ενώ το τρίτο μήνυμα είναι κάποια, κάποιες προτάσεις για την βελτίωση θέμα, του θέματος ασφάλειας δικαίου για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, μια κατάσταση των πραγμάτων, μια γενική επισκόπηση. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πολύ διαφορετικέ καταστάσει. Μόνο πέντε χώρε μέλη αναγνωρίζουν το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Η Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, κατοχώρε και Βέλγιο. Άλλε χώρε αναγνωρίζουν ε, συμφωνίε συμβίωση, αλλά για ομοφυλόφιλους που ουσιαστικά όμως ε, είναι πιστή αντιγραφή του γάμου αλλά με τη μορφή συμφωνίας συμβίωσης. Άλλες χώρες, ε, αυτό ισχύει για τη Γερμανία, τη Δανία για παράδειγμα, άλλες χώρες αναγνωρίζουν συμφωνίες ε, συμβίωσης που είναι κάτι σαν συμβόλαια, κάποιες συμβάσεις ουσιαστικά που προσφέρονται κυρίως προσφέρονται και σε ομοφιλόφιλα και σε τεροφιλόφιλα ζευγάρια, είναι ανοιχτά προς όλους δηλαδή, αλλά έχουν πολύ ασήμαντα νόμα αποτελέσματα. Χώρε όπως η Πολωνία και άλλες χώρες δεν αναγνωρίζουν ούτε το γάμο μεταξύ ομοφιλοφίλων ούτε τη συμφωνία συμβίωση. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά. Δηλαδή κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορά ε, με διαφορετικό τρόπο τις, ε, τους γάμους που γίνονται σε άλλες χώρες. Γιατί ε, κάτι που χαρακτηρίζεται γάμο σε μια χώρα, σε άλλη χώρα μπορεί απλώς να χαρακτηρίζεται συμφωνία συμβίωσης. Επίσης ισχύουν διαφορετικές ε, νομοθεσίες και νομοθετικές διατάξεις για τις άνομες συνέπειες αυτών των ε, ενώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμοστέο δίκαιο είναι της υπηκότητας, ε, της διαμονής ή της, της χώρας της σύναψης του γάμου. Επίσης άλλε χώρες για λόγους δημόσιου αντιστέκονται στην αναγνώριση του γάμου ομοφιλοφίλων. Μεγάλη αταξία δηλαδή και μεγάλες διαφορές. Ας πάρουμε το παράδειγμα ενό Γάλλου και ενός Ισπανού ομοφιλόφιλου που παντρεύονται στην Ισπανία. Αυτός ο γάμος είναι έγκυρος και ισχύει στην Ισπανία, αλλά είναι ανυπόστατο άκυρο στη Γαλλία. Μία πρόσφατη δικαστική απόφαση Γερμανικού Δικαστηρίου θεώρησε ότι γάμος μεταξύ ομοφιλοφίλων μόνο σε συμφωνία συμβίωσης μπορεί να αναγνωριστεί στη Γερμανία. Η, μόνη, η νόμιμη συμβίωση στο Βέλγιο μεταξύ ε, διαφορετικών φίλων ανθρώπου δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια συμφωνία συμβίωση στη Φιλανδία, γιατί στη Φιλανδία επιτρέπονται τη συμφωνία συμβίωση μόνο μεταξύ ομοφιλοφίλων θα πρέπει να χαρακτηριστεί με διαφορετικό τρόπο, είτε γάμος είτε ως de facto συγκατοίκηση, συμβίωση. Ενώ μια νόμιμη συμβίωση στο Βέλγιο μεταξύ δύο ομοφυλοφίλων αναγνωρίζεται ε, κάλλιστα ως ε, τέτοια και στη Φιλανδία. Μια γερμανική συμφωνία συμβίωσης που έχει κυκλονομικές συνέπειες για τη Γερμανία δεν αναγνωρίζεται στη Γαλλία για παράδειγμα μία δευτερεύουσα κατοικία που αγοράζουν δανείς στη Γαλλία, δεν ξέρω ε, σε τι εφαρμοστέο δίκαιο θα υποπέσει για το καθεστώς αυτό των περιουσιακών στοιχείων της δοσιδικίας του δικαστηρίου, της, ε, του χώρου, του, του τόπου του αγαθού ή της καταγωγής του ιδιοκτήτη. Υπάρχουν πολλές διαφορές Έχουμε βέβαια ελευθερία κυκλοφορία, αλλά δεν υπάρχει σχετική νομολογία του ΔΕΚ για τέτοιου είδου ζητήματα. Έχουμε νομολογία ως προς το ο... όνομα που ισχύει όταν αναγνωρίστε σε ένα κράτος και στα υπόλοιπα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο και τις ενώσεις. Το δικαίωμα της οδηγίας του 2004 προβλέπει ότι ένας σύντροφος μπορεί να θεωρηθεί ο σύζυγος αν η συμφωνία συμβίωση έχει τέτοια αποτελέσματα και τις ένωμες συνέπειες με το γάμο. Έχουμε το άρθρο, το άρθρο 12, το άρθρο 8, το άρθρο 14 των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εκεί Μιλούμε για το δικαίωμα γάμου, σεβασμό τη ε, οικογενειακή ζωή και απαγόρευση διακρίσεων για λόγου προς ανατολισμού. Δεν έχουμε όμω νομολογία του ΔΕΚ, ε, ούτε μάλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ομοφυλόφιλε σχέσει, ε, για ομοφυλόφιλε ενώσει. Μόνο μία αυστριακή απόφαση επιτρέπει πρόσφατα τα κράτη-μέλη να αρνηθούν να εγγράψουν ή να κατοχυρώσουν το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων στην ομοθεσία του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εφαρμόσει νομολογία για την αναγνώριση κάποιων καταστάσεων που δημιουργούνται στο εξωτερικό, όπω η οθεσία. Απόφαση Λουξεμβουριανή Δικαστηρίου, ή μάλλον κατά του Λουξεμβούργου, ή απόφαση διασγείου κατά τη Τουρκία. Έχουμε όμω το άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που προβλέπει ότι έχουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε οικογένεια, αλλά αυτό το δικαίωμα κατοχυρώνεται από το εθνικό δίκαιο. Μεγάλη αβεβαιότητα δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το διεθνέ δίκαιο, ούτε και εκεί υπάρχει νομολογία, γιατί το θέμα είναι πολύ πρόσφατο και η θεωρία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν διστάμενε απόψεις. Μερικέ φορέ πριτανεύει το δίκαιο προέλευση για τις συμφωνίε συμβίωση. Άλλοι μιλούν για το τοπικό δίκαιο που εξομοιώνεται με το δίκαιο της προέλευσης. Τεράστια νομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα λοιπόν. Για να βάλουμε μια τάξη σε όλα αυτά, ποιες λύσεις υπάρχουν. Είτε θα μπορούσαμε να ενοποιήσουμε το ουσιαστικό δίκαιο, αλλά αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, είτε να ενοποιήσουμε τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Υπάρχουν κάποιες καλές πρωτοβουλίες, αλλά βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της περιπέτειας. Ίσως θα δούμε, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει πριν ανοίξουμε νέα μέτωπα. Επίσης θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε πιο μετριοπαθείς λύσεις. Για παράδειγμα, την αναγνώριση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αναγνώριση των αλλοδαπών ενώσεων με το χαρακτηρισμό της χώρας στην οποία συνάπτονται. Και κάτι άλλο πιο φιλόδοξο, μπορούμε να δώσουμε έμφαση στον κανόνα συνάφειας αιτιών και αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι μία ένωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη με το χαρακτηρισμό του κανόνα προέλευσης, ε, φυσικά αποκλείοντας τις περιπτώσεις απάτης Δηλαδή, ένας γάμος μεταξύ μεταξύ ομοφυλόφιων Σουηδών να χαρακτηρίζεται παντού γάμος και όχι σε ορισμένε χώρες συμφωνία συμβίωση. Ένα γαλλικό παξ, να παραμένει παξ, ακόμη και αν α, οι σύντροφοι μένουν στην Φιλανδία, για παράδειγμα. Έτσι θα μπορούν οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μπορούν να συνάπτουν τις ενώσεις, τους γάμους, τις συμφωνίες συμβίωσης, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Υπάρχουν αποσπασματικές διατάξεις, για παράδειγμα μιλήσαμε για τις υποχρεώσεις διατροφής, για το διαζύγιο, για τις κληρονομικές σχέσεις, κληρονομικές διατάξεις, για το καθεστώς περιουσιακών σχέσεων, επίσης για φορολογικά ζητήματα υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια της σύνδεσης των κανόνων, ρατασμό, για παράδειγμα, να συνδέεται η συμφωνία σύνδεσης με τον νόμο του, τόπου καταγραφής αυτής της συμφωνίας καλύτερο θα ήταν να αφήσουμε τους συζύγους ή τους συντρόφους να διαλέγουν το εφαρμοστό δίκτυο. δίκτυο. Τι μπορεί να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα είναι να επιτρέπει αυτή την αναγνώριση. Χρειαζόμαστε όμως ένα μηχανισμό που θα επιβάλλει στα κράτη-μέλη αυτή την αναγνώριση με τον αρχικό της χαρακτηρισμό, τον αρχικό χαρακτηρισμό όλων αυτών των ενώσεων. Είναι πολύ ευαίσθητο και λεπτό το θέμα του ορισμού που μας προβληματίζει πολύ συχνά στην νομοθεσία. Ποια είναι η συνήθις κατοικία, να, να καθορίσουμε υπό ευρωπαϊκή έννοια μια συνήθεια κατοικία. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Επίση θα πρέπει να ορίσουμε με ευρωπαϊκό τρόπο το γάμο ή τη συμφωνία συμβίωση. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, τις ένομες συνέπειες, νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύσουν ε, συνθήκες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και να δώσουμε έμφαση στη σύγκληση μεταξύ των διαφόρων διατάξεων, παροτρύνοντας τις χώρες να σεβαστούν τη φύση τη συγκεκριμένη ένωση όταν εφαρμόζουν το δίκαιό τους για τις ένομε συνέπειε μια τέτοια ένωσης ή συμφωνία συμβίωση. Για την αναγνώριση υπάρχει αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων για παράδειγμα. Από τη στιγμή που μια ένωση συνάπτεται ή εορτάζεται ή γίνεται μπροστά σε μια δημόσια αρχή, το θέμα της αναγνώρισης νομίζω είναι στοιχειώδες είναι αυτό που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χώρα για να σεβαστεί την νομοθεσία άλλης χώρας μέλους. Επίση θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσει αλλοδαπό δίκαιο. Γιατί στη τελική ανάλυση, συμφωνώ με την κυρία Μπέκερ, νομίζω ότι δεν θα έχουμε Ευρώπη αν δεν φέρουμε πιο κοντά τις νομοθεσίε μα και την αντίληψη που έχουμε για το δίκαιο και την κατανόηση και του αλλοδαπού δικαίου. Είναι σημαντικό όλοι να γνωρίζουμε και τις ε, νομοθετικές διατάξεις των άλλων χωρών. Έτσι θα εμπλουτιστεί ο διάλογος μεταξύ μας και θα γίνει ένα είδος προσέγγισης ε, όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα αλλά και ε, από μέρους της νομικής και της δικαστικής κοινότητας. Και έτσι αναλαμβάνουμε και εμείς ένα τμήμα της ευθύνης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και πολύ ενδιαφέρουσες και ακριβέστατες οι προτάσεις σας. Βέβαια για μερικούς είναι δύσκολη αποδοχή τέτοιων προτάσεων και θυμάμαι συζητήσεις που είχαμε σχετικά στην ε, Ολομέλεια. Πάντως ήταν πραγματικά μονοσήμαντες οι προτάσεις σας, κατηγορηματικές, αφέστατες, ξεκάθαρες και σίγουρα θα μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν τροφή στη συζήτηση. Ο επόμενος εμπειρογνώμονας σε αυτό το τμήμα είναι ο κύριος Τσάρλς Χάιτ, ε, μπαριστερ, δικηγόρος, ε, μέλος του Δικαστικού Συλλόγου του Λονδίνου. Is that Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι Άγγλος και μου αρέσει το roast beef. Δεν ξέρω, δεν ξέρω γαλλικά καλά, δεν ξέρω καθόλου φλαμανδικά ε, και μέχρι 18 χρονών δεν ήξερα τι συμβαίνει έξω από την Αγγλία. Ε, είχα πάει μέχρι τη Σκωτία όμως και χρησιμοποίησα τη Σκωτία σαν τόπο διαφυγής από την ε, Αγγλία. Για, όταν ήμουν 18 χρονών έφυγα πρώτη φορά λοιπόν, πήγα στο εξωτερικό τότε για πρώτη φορά, πήγα στην ε, Αυστραλία γιατί μιλάνε αγγλικά εκεί. <laughs> Και ίσως είναι περίεργο που μου ε, ζητήθηκε ε, να σας δώσω την άποψη του ε, βρετανικού δικαίου για το θέμα αυτό. Ξέρετε, στην Αγγλία είμαστε πολύ παραδοσιακοί Είμαστε και πολύ πεισματάριδες και δεν είμαστε και εύκολοι, ούτε παίρνουμε εύκολα αποφάσεις και γρήγορα. Και ενδεχομένως αυτά που θα σας πω σας φανούν προοδευτικά ή βολικά, αλλά θα, θα ήθελα να σας πω ποια είναι η άποψή μας όσον αφορά την, ε, τον γάμο και τις ε, ενώσεις ε, ομοφύλων. Από τη Βικτωριανή εποχή έχει ξεκινήσει η διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες από τη Βικτωριανή εποχή δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφους, ψήφου μια γυναίκα που παντρευόταν στη Βικτωριανή εποχή δεν είχε πλέον κανένα δικαίωμα. Ο άντρα ήταν αυτό ο οποίο ε, ε, ε, είχε πλήρη κυριότητα κατά κάποιο τρόπο πάνω στη γυναίκα και τα παιδιά της και την περιουσία της. Και βεβαίως η γυναίκα δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποφασίσει ότι θέλει να διαλύσει το γάμο. Το 1973 στην ουσία άλλαξαν κάποια πράγματα και από τότε καμία άλλη. 37 χρόνια έχουμε ε, νομική ερμηνεία του αρχικού νόμου και αυτό είναι ακόμα πιο εμφανές όταν ε, αναφερόμαστε στα οικονομικά δικαιώματα ε, μέσω ενός συστήματος μη αντικειμενικού καταμερισμού. Ε, ενδεχομένως ε, ο νόμος εξακολουθεί ε, να είναι προβληματικός όσον αφορά τις γυναίκες και όντως ήταν μέχρι το 2000. Το 2000 λοιπόν ορίστηκε μια, ένα μια οροφή όσον αφορά ε, τις απαιτήσεις ε, που μπορούσαν να έχουν ε, οι γυναίκες. Και λίγο αργότερα το δικαστήριο αναγνώρισε ότι δεν υπήρξε αντικειμενικό στις οικονομικές εκτιμήσεις του μέχρι τότε. Είχαν μερικοί την εντύπωση ότι ε, ο αρχικός νόμος ήταν καλύτερος. Στην ουσία δεν ήταν καλύτερος όμως. Ήδη από το 1954 ζητήθηκε από τον Λόρδο Βόλφ ε, να κάνει μία έρευνα ε, όσον αφορά τους, ε, την σεξουαλικότητα και όσον αφορά την δυνατότητα φυλάκισης για σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ μεταξύ ε, Μετά την έρευνα αυτή ε, αποφασίστηκε ότι δεν μπορούσε να αποτελέσει αιτία εγκλισμού ε, τέτοιου είδους σεξουαλική επιλογή. Στη Σκωτία τα πράγματα άλλαξαν με πολύ αργότερο ρυθμό. Το 2002 οι ε, ομοφιλόφιλοι άνδρες ε, ε, είχαν πλέον το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά και δύο χρόνια αργότερα είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν γάμο. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί οι αλλαγές που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία είναι τρομερές όχι μόνο το ε, ημεδαπό δίκαιο έχει τροποποιηθεί, αλλά, και αυτό είναι πιο σημαντικό, έχει υπάρξει αναγνώριση ε, των ε, δικαίων των λοιπών χωρών της Ευρώπης. Γίνεται αποδεκτή γίνονται αποδεκτά τα δικαιώματα τα οποία εμπεριέχονται σε μία σχέση και οι υποχρεώσεις ανεξαρτήτως τι είδους σχέση είναι αυτή και μπορεί κανείς πλέον να ε, ξεκινήσει διαδικασία γάμου ε, ακόμα και αν πρόκειται για άτομα του ιδίου φύλου. Ε, αυτό δεν ισχύει βεβαίω μονάχα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, και, αλλά και σε άλλες χώρες. Ε, ε προβλέπονται επίσης πέραν του γάμου και κάποιες εταιρικές αστικές σχέσεις και επομένως αναγνωρίζονται και τέτοιου είδους σχέσεις που έχουν προκύψει σε άλλες χώρες του κόσμου βεβαίως λαμβάνοντας ε, υπόψη κάποιες προϋποθέσεις ε, και κάποιους ε, όρους. Τα λαμβάνονται φυσικά υπόψη και τα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται ε, στο ε, ζευγάρι από, άλλη, από κάποιο άλλο δίκαιο. Ε, δηλαδή, εάν το ζευγάρι έχει παντρευτεί σε μια άλλη χώρα, στην Μεγάλη Βρετανία θα αναγνωριστούν τα δικαιώματα, ακόμα και αν πρόκειται για υλικά δικαιώματα και για αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για το διαζύγιο. Και εάν η λύση του γάμου έχει λάβει χώρα σε άλλη ε, χώρα ε, παρόλα αυτά το εν λόγω ζεύγος μπορεί να ζητήσει ε, τον καταμερισμό της περιουσίας και των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού στην Μεγάλη Βρετανία. Το ίδιο ισχύει και εάν πρόκειται για δεσμό που δεν είναι γάμος. Εάν όμως υπάρχουν παιδιά, η γονική μέρημνα δίνεται ε, στο, στον σύζυγο εάν το όνομά του αναφέρεται εις το πιστοποιητικό γέννησης. Το, 1990 αναφέρθηκαν για πρώτη φορά και τα δικαιώματα των μη βιολογικών γονέων καθώς επίσης και των γονέων παιδιών που έχουν προκύψει από παρένθετες μητέρες ή από But it has to deal with another dimension. από διαδικασίες τεχνητής ε, γονιμοποίησης ε, in vitro. Ε, αναγνωρίζονται επίσης δικαιώματα στην φέρουσα μητέρα. Βεβαίως ε, δεν ε, ε, υπάρχει αναδρομική ισχύς για τους γονείς, μη βιολογικούς γονείς που όμως ζουν σε ελεύθερη σχέση και όχι με κάποια, μέσα σε κάποια σχέση καταγεγραμμένη. Το ημεδαπό δίκαιο μας έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε ε, όταν ε, υπάρχει γονική μέρημνα η οποία έχει αναγνωριστεί σε άλλη χώρα ε, ακολούθως να αναγνωρίζεται και στη δική μας χώρα. Και κατά την άποψή μου αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που έχω να σας μεταφέρω. Η αναγνώριση στο ημεδαπό δίκαιο της νομολογίας άλλων κρατών αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εναρμόνισης του δικαίου, έστω και αν δεν υπάρχει ομοιογένεια δικαίου. Δουλέψαμε πάρα πολύ κατά την άποψή μου, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε και να εφαρμόσουμε το δικαϊκό σύστημα ε, των άλλων χωρών. Σεβόμαστε την ε, νομολογία των άλλων ε, χωρών και ε, ε, το ε, δίκαιο διαζυγίου πιστεύουμε ότι πλέον μπορεί να εξαχθεί και σε άλλες χώρες και να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες ικανοποιητικά. Ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί τα μάλα και από το ρυθμό αλλά και από το περιεχόμενο των αλλαγών και των τεράστιων μεταρρυθμίσεων στο Βρετανικό Δίκαιο σε ό,τι αφορά το γαμικό δίκαιο και το οικογενειακό δίκαιο και σας ευχαριστώ και για τα συμπεράσματά σας. Δυστυχώς ε, ο χρόνος τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη δυνατότητα που έχετε να λάβετε μέρος στη συζήτηση που θα αρχίσει εδώ σε λίγο. Παρακαλώ δηλώστε ενδιαφέρον συμμετοχής για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε και τη συζήτηση. Το τελευταίο θέμα του πάνελ αυτού είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και ουσιαώδες θέμα σε ό,τι αφορά την προστασία της οικογένειας, αλλά ιδιαίτερα των παιδιών, που είναι τα πιο ευάλωτα στοιχεία αυτής της οικογένειας. Θα δούμε τι κατάσταση επίκρατη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας την παρουσιάσει η κυρία Μαρία Ντακοσεϊσάου Ολιβέηρα, που είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής από την Πορτογαλία και εμπειρογνώμονα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχετε το λόγο κυρία Μαρία Ολιβέρα. Ε, Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ και Βουλευτέ. Η διεθνής ε, μεσολάβηση σε οικογενειακά ζητήματα αναπτύχθηκε πολύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες χάρη σε πολλές και διάφορες πρωτοβουλίες. Αυτή η πρόοδος δεν οφείλεται μόνο στην πρόθεση των ε, κυβερνήσεων και των ε, αρμοδίων αρχών, αλλά και στη συμμετοχή των δικαστικών νομομαθών, ψυχολόγων, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για ένα φιλικό, εμπιστευτικό διακανονισμό που θα σέβεται και τα δύο συμβαλόμενα μέρη στη σύγκρουση συμφερόντων. Στο θέμα του οικογενειακού δικαίου η μεσολάβηση είναι από τους πιο γνωστούς εξώδικους ε, τρόπους διευθέτησης διαφορών, ακόμη και σε θέματα διαζυγίου, σε θέματα γονικής μέρημνας. Μερικές φορές ε, οι συγκρούσεις ε, είναι τόσο ακραίες που οδηγούν ακόμη και σε απαγωγή των παιδιών από τον ίδιο το γονέα. Είναι σημαντικά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης γιατί λαμβάνει υπόψη τις ε, ψυχολογικές συνέπειες των ε, οικογενειακών συγκρούσεων για όλους τους ε, εμπλεκόμενους. Και η διαδικασία της διαμεσολάβησης, η βοήθεια του διαμεσολαβητή προς, τα, προς αντιδίκους εξασφαλίζει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας που είναι προς όφελος των παιδιών και λαμβάνει υπόψη και το μέλλον και τις ιδιαιτερότητες φυσικά. Φυσικά, ο καλύτερος ε, γνώστης των αναγκών των παιδιών είναι οι γονείς τους. Και παρά το διαζύγιο υπάρχει δυνατότητα διαμεσολάβησης. Χάρη στη διαμεσολάβηση ε, έχουμε μια λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση από ότι με την άσκηση αγωγής και τη δικαστική απόφαση. Ε, βέβαια, με τη επίσημη τη διαμεσολάβηση, ακριβώς επειδή είναι φιλικός ο διακονονισμός και η παράβαση των υποχρεώσεων είναι πιο σπάνια. Στην Ευρώπη η διαμεσολάβηση προσπαθεί να δώσει απάντηση σε δύο σημαντικές ανησυχίες. Την ανάγκη προστασίας των παιδιών αφενός, αλλά και την συμπλήρωση της δικαστικής αποτελεσματικότητας. Στηριζόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία, στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Γι' αυτό και η διαμεσολάβηση εκεί διαδραματεί σημαντικό ρόλο. Έχουμε τη σύσταση για την οικογενειακή διαμεσολάβηση του 1998. Ήταν πολύ σημαντικό εργαλείο και αποτέλεσε τον πρόδρομο σημαντικών πρωτοβουλειών. Πρόσφατα είχαμε τις κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δικαστική αποτελεσματικότητα το 2007. Αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές βοηθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις για θέματα διαμεσολάβησης, όχι μόνο για οικογενειακά ζητήματα, αλλά και για άλλα θέματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Οδηγία 2008 για διάφορα θέματα διαμεσολάβησης σε εμπορικά και αστικά ζητήματα ε, συνοδεύτηκε και από άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η δικαστική αρρωγή και σε θέματα εξώδικης ο οδηγία του 2003, ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α που προσφέρει δυνατότητα δικαστικής διατησίας. Έχουμε και την έκθεση για τις διάφορες δικαστικές πτυχές, τις στατιστικές του 2008 και χάρη σε αυτή την πρόσφατη έκθεση αναγνωρίζεται η σημασία της διαμεσολάβησης, ιδιαίτερα για οικογενειακά ζητήματα που και μάλιστα παρα, παρατηρούμε μία ανωδική τάση στην Ευρώπη. Ο ρυθμός των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών όλο και αυξάνεται. Και αυτό φυσικά εννοείται στι χώρε όπου υπάρχει τέτοια διαπίστευση κατά κάποιο τρόπο διαμεσολαβητών. Υπάρχει εξουσιοδότηση συγκεκριμένων διαμεσολαβητών. Εκεί έχουμε τέτοια στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση, δυστυχώ εκεί η εικόνα δεν είναι τόσο θετική. Παρόλο που αναγνωρίζεται η ανάγκη τη για τι διασυνοριακέ ε, συγκρούσεις ε, με βάση στοιχεία που έχουμε από το 2003, αρκετά παλιά. Το 2003 το 17% των διαζυγίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διασυνοριακή διάσταση, διακρατικό χαρακτήρα. Και μάλιστα Έχουμε πολλέ οικογενειακέ αντιδικίε που έχουν μια τέτοια διασυνοριακή διάσταση. Αυτέ οι αντιδικίε μένουν πολλέ φορέ χωρί λύση, γιατί το δικαστικό σύστημα έχει προβλήματα και πολλού περιορισμού που εμποδίζουν την άμεση διευθέτηση των οικογενειακών διαφορών. Παρά τα προσκόμματα όμως που εμποδίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη της διαμεσολάβησης σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η έλλειψη κρατικών δημόσιων πρωτοβουλειών, η εξασφάλιση ποιότητας ε, υπηρεσιών, η εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Υπάρχουν και άλλα εμπόδια, πολύ συγκεκριμένα, για την διεθνή οικογενειακή μεσολάβηση. Για παράδειγμα, νομοθετικές διαφορές, δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών, γεωγραφικοί παράγοντες, αλλά και πολιτιστικές διαφορές. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα ανυπέρβλητα κάποιες φορές για τη διαμεσολάβηση. Η οικογενειακή διεθνή διαμεσολάβηση είναι και μια ειδίκευση. Είναι μια ειδίκευση που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή ένας οικογενειακός διαμεσολαβητή μπορεί να έχει διάθεση να ασχοληθεί με τη διεθνή οικογενειακή μεσολάβηση, αλλά για να το κάνει θα πρέπει να διαθέτει και άλλες αρμοδιότητες και άλλα προσόντα και άλλα εφόδια που είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια επιμόρφωση, τέτοια κατάρτιση για οικογενειακή διαμεσολάβηση. Γνωρίζουμε ότι στο Βέλγιο βρίσκεται στα σπάργανα μια τέτοια κατάρτιση για διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση, αλλά επαναλαμβάνω βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ πρωτόλια φάση αυτής της διαδικασίας. Η προθεσμία για την ε, μετάθεση της οδηγίας του 2008 για τη μεσολάβηση θα λήξει το Μάιο του 2011. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι κάπως πρόωρο να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις ε, για την επίπτωση που θα έχει εφαρμογή αυτή τη οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Βέβαια, οι διαμεσολαβητές είμαστε της γνώμης ότι η οδηγία αυτή θα δώσει μια θαυμάσια ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της διαμεσολάβησης και όχι μόνο της διασυνοριακής διαμεσολάβησης που κατοχυρώνει η οδηγία, αλλά και η διαμεσολάβηση εντός των χωρών μελών, η εσωτερική διαμεσολάβηση θα αναπτυχθεί χάρη στην οδηγία. Γιατί η οδηγία και η μετάθεσή της στο εσωτερικό δίκαιο θα επιτρέψει την διαμόρφωση προϋποθέσεων για την διαφκόληση της οικογενειακής διαμεσολάβησης και σε εσωτερικές ε, διαφορές οικογενειακές. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή τώρα οικογενειακή διαμεσολάβηση, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό α, την εξετάσουμε με διαφορετικό πρίσμα και να επενδύσουμε κυρίως σε τρει διαφορετικούς τομείς. Στον τομέα τη ειδικευμένη επιμόρφωσης και κατάρτιση και εναρμονισμένης για την διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση, που ίσω οδηγήσει στη δημιουργία ενό διπλώματο ή ενό ευρωπαϊκού πιστοποιητικού του οικογενειακού διεθνούς διαμεσολαβητή. Επίσης θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση στην ε, αφύπνιση των δικαστών ή των νομικών. Θα μπορούσαμε να δίνουμε τέτοιες συμβουλές ε, στους αντιδίκους ε, να προτιμούν έναν εξώδικο διακανονισμό, μια διαμεσολάβηση. Και είναι σημαντική εδώ η ευαισθητοποίηση των δικαστικών αρχών και των νομικών. Φυσικά η διαμεσολάβηση δεν είναι πανάκια, αλλά σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση είναι κατάλληλη, ένας δικηγόρος που είναι κοντά στους πελάτες ε, θα μπορούσε να τους ευαισθητοποιήσει ως προς αυτή την κατεύθυνση και ο ίδιος να είναι ευαισθητοποιημένος. Να γνωρίζουν καταρχήν οι άνθρωποι ότι υπάρχει δυνατότητα του, της διαμεσολάβησης. Εγώ Είμαι μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστών υπέρ της διαμεσολάβησης, γιατί και αυτό το δίκτυο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη αυτού του σημαντικού μέσου διακανονισμού των διαφορών. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε μεγαλύτερη δέσμευση και ενθουσιασμό τα κράτη-μέλη στην ε, διάδοση και την υποστήριξη της διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης. Να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτή, ακόμη και όταν ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν ε, τα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσουν ε, τα έξοδα αυτής της διαμεσολάβησης, που όταν έχει διεθνή χαρακτήρα είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι ήταν εσωτερική διαμεσολάβηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό πλαίσια των πολύμορφων και πολυπολιτισμικών κοινωνιών μας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι αυτή η πολυμορφία και νομίζω ότι θα πρέπει να την υποστηρίξουμε και να την προωθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Ολιβέρα. Ευχαριστώ θερμά όλους του εμπειρογνώμονε μας, όλους τους πανελίστε, για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσε παρουσιάσεις του και επί της ουσίας αλλά και επί του τύπου γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από την αυστηρή τήρηση του χρόνου. Φάνηκε από, την, ε, από τις παρουσιάσεις αυτές ότι όταν κάποιος έχει ένα, ένα πολύ σημαντικό και μεστό μήνυμα να διαβάσει μπορεί να το κάνει και σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν είναι σαφής. Ωραία, προχωρούμε τώρα στη συζήτηση. Δύο ε, εθελοντές ζήτησαν το λόγο. Κάτι που θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε εγκαίρως το δικό μας πάνελ και θα δώσω το λόγο στο τέλος ένα πεντάλεπτο περίπου στο γερουσιαστή για να κάνει μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε από ό,τι φαίνεται 15 20 λεπτά για την ανταλλαγή απόψεων. Το λόγο ζήτησε πρώτα ο κύριος Στέφαν Πρόμε από το γερμανικό Bundestag. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εν ονόματι της Γερμανικής Βουλής σας ευχαριστώ για την εργασία και τη συζήτηση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας καλέσατε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ομιλητή που έθιξε το θέμα της ε, τρίτης συμβάσεως της Ρώμης. Ε, ήταν μια εξαιρετική ε, ομιλία παρόλο που κυρία και πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν συμφωνώ πλήρως μαζί σας και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εδώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν το τελευταίο κοινό ο τελευταίος κοινός χώρος διαβίωσης του ζευγαριού πρέπει να είναι αποφασιστικός για τις διαδικασίες του ε, διαζυγίου διότι υπάρχουν καλοί λόγοι ε, για να θεωρήσει κανείς ότι θα πρέπει κανείς να αναφερθεί εις το σημείο όπου έζησαν από κοινού μαζί οι σύζυγοι ε, τελευταία πρώτου διαζυγίου ακόμη και αν έχουν φύγει από το σημείο αυτό τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση διαζυγίου διότι ε, πρέπει κανείς να ε, σκεφτεί ότι ίσως οι διάδικοι έχουν διαβιώσει σε ένα ουδέτερο δίκαιο και αυτό το ουσιαστικό δίκαιο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ε, στην περίπτωση αυτή και όπως σας είπα και προηγουμένως έτσι ε, αναφέρεται κανείς στα κοινά σημεία κατά τη διάρκεια της συζυγικής ζωής ε, ακόμη και αν λοιπόν οι σύζυγοι δεν διαβιούν πλέον στο σημείο αυτό και αυτό ρυθμίζεται στο σημείο 3 της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3.1 ένα β όπου λέγεται ότι ε, θα λυθεί η διαφορά στο τελευταίο σημείο που διαβίωσαν οι σύζυγοι ε, αρκεί κάποιος από τους δύο να διαβεί ακόμη εκεί και εγώ θα σας έλεγα περαιτέρω ότι ακόμη και αν δεν μένει κανείς από τους δύο σύζυγους πλέον εκεί ακόμη και τότε ε, μπορεί να διαλέξει κανείς το δικαίωμα του, το δίκαιο του κράτους όπου ε, έμεναν ε, οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου επί πολύ χρονικό διάστημα. Ίσως θα έπρεπε αυτό να αναφερθεί και με αυτό θα ήθελα να συνδυάσω μία ε, ερώτηση σχετικά με το ουσιαστικό δίκαιο, σχετικά με την δικαιοδοσία. Δηλαδή, μήπως θα πρέπει να επιλεγεί η δικαιοδοσία του χώρου που έζησαν από κοινού ακόμη και αν κανένας από τους δύο δεν έχει πλέον στο κράτος αυτό τη συνήθη διαμονή του διότι αυτό ήταν ένα σημείο όπου είχαν συνδεθεί και οι δύο κατά τη διάρκεια του γάμου. Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στη συνέχεια, να κάνω μια σύντομη παρατήρηση, γιατί είμαι εισηγητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Συμφωνώ μαζί σας για τον τόπο, για τον τελευταίο τόπο κοινή συμβίωσης κατοικία, αλλά ο κανονισμός Ρώμη 3 αφορά την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, όχι την, την επιλογή της ε, δικαιοδοσίας ή ειδικία. Μια σημαντική νομίζω διευκρίνηση αυτή. Äh, Ευχαριστώ. Η παρατήρηση του Προέδρου είναι πολύ σωστή, διότι θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο ε, τελευταίο θέμα, διότι η επιλογή της ε, ε, δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην συνθήκη Βρυξέλλες 2 και αυτό υπήρχε στο αρχικό σχέδιο το 1988. Ελπίζουμε όμως ότι στο μέλλον θα είναι δυνατόν και αυτό να καλυφθεί, όχι όμως στον ε, κανονισμό αυτό. Λογικά δεν μπορεί να ρυθμιστεί τώρα. Όσον αφορά την τον συνήθι τόπο διαβίεσης εις ε, την ε, συζήτηση για, που έγινε στην Ολλανδία για ένα ένα ε, ε, διεθνές δίκαιο ως προς τα διαζύγια πολύ σωστά ελέγχθη ότι το σημείο αυτό είναι περίπλοκο διότι πρέπει εκ των υστέρων να ε, διαπιστωθεί ιδίω όταν πρόκειται για επιλογή ισχύοντος δικαίου οπότε αυτό δεν πρέπει να ισχύσει ίσως μόνο τη στιγμή του διαζυγίου αλλά και στην αρχή του γάμου ή κατά τη διάρκεια του γάμου και ε, αυτό το δικαίωμα χρησιμοποιείται για να διαπιστώσει κανείς ε, τον, ε, το κοινό σύνηθε σημείο διαβίωσης κατά τη διάρκεια του γάμου. Οπότε το Lex το δίκαιο το οποίο επιλέγεται είναι πολύ πιο εύκολο να επιλεγεί εάν μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες ε, άλλες ε, συνθήκες ε, και διάφορα χαρακτηριστικά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο απέθυναν παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να κάνει σύντομη αναθεώρηση και να υποβάλει προτάσεις ε, μεταρρύθμισης ε, της πρότασης Βρυξέλλες 2α. Ε, Νομίζω ότι αναμένεται αναθεώρηση. Δεν περιμένω καμία επανάσταση, άλλως αυτό θα γίνει το συντομότερο το 2003 εκτός και αν ληφθούν υπόψη οι πιέσεις μας και οι κλήσεις μας για επίσπευση των εργασιών, αλλά ίσως για αυτό θα μπορούσε να μας απαντήσει η αρμόδια επίτροπος, η κυρία Ρέντινγκ. Επόμενος ο μιλητής μας είναι ο γερουσιαστής Σενάρ Γιούγκ από την Γαλλική Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους ε, οργανωτές αυτής της ε, ε, ημερίδας. Πρόκειται για εξαιρετικά επικοδομητική ημερίδα ε, και πολύ ενημερωτική για ανθρώπους που ενδεχομένως ε, δεν είναι τόσο γνώστες του αντικειμένου ε, και που όμως πρέπει να συζητήσουν τα θέματα αυτά στα εθνικά τους κοινοβούλια. Πρόκειται βεβαίως και για ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο γιατί αντίστοιχα και με την εκπαίδευση, ε, αγγίζοντας τα θέματα αυτά, αγγίζουμε τη βάση της κοινωνίας, τη βάση επί της οποίας οικοδομείται η κάθε χώρα. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι πρόκειται για θέματα εξαιρετικά περίπλοκα ε, ακροβατούμε μεταξύ Ρώμης 3, Βρυξέλλες 1, Βρυξέλλες 1α ε, κλπ. Ε, και προσπαθούμε να βρούμε ένα μπούσουλα για να ξέρουμε προς τα που θα προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά αυτή η διαλεκτική συζήτηση που έχει ξεκινήσει είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες πιθανές οδούς που μπορεί να ακολουθήσει κανείς έτσι ώστε να προωθήσει τα πράγματα ε, και αυτό μας ε, ικανοποιεί. Ε, υπάρχει η δυνατότητα της διευρυμένης συνεργασίας και κατά την άποψή μου ε, αυτό είναι σημαντικό ε, και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να αναλυθούν και σε άλλους τομείς και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και ε, διμερείς πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες και λύσεις μεταξύ δύο κρατών ας πούμε το έχουμε δει στην περίπτωση των γαλλογερμανικών σχέσεων που καταδεικνύει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και με δύο και με τρεις και με τέσσερις και σιγά σιγά να φτάσουμε στους 20 27. Επομένως ε, μπορούμε να βρούμε 27 τρόπους να προχωρήσουμε ε, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και πιστεύω ότι είναι καλό. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Εύα Μπέκερ που μας ε, εξήγησε το γαλλογερμανικό γαμικό καθεστώς. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές, ε, ε, πολλά, πολλοί γαλλογερμανικοί γάμοι και επομένως ε, υπάρχουν αρκετές συγκρούσεις όσον αφορά τα θέματα αυτά και για τα διαζύγια και για την μέρημνα των παιδιών κλπ. Και βεβαίως Ξέρουμε ότι το πρόβλημα δεν, είναι, δεν προκύπτει μονάχα από παιδιά που έχουν προκύψει από γαλλογερμανικούς ε, γάμους. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ε, όσον αφορά γάμους μεταξύ Ευρωπαίων και Ιαπώνων και μεικτά ζευγάρια που εκεί σε περίπτωση διαζυγίων έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και ασχολούμαστε με το θέμα αυτό στην Γαλλική Γερουσία. Βεβαίως ε, ξεφεύγει από την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ε, ε, συμφωνία, η γαλλογερμανική ε, συμφωνία για το γάμο και ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί να συμμετάσχουν στην συμφωνία αυτή, αλλά ακόμα είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η, τώρα ένα άλλο ζήτημα, η αμοιβαία αναγνώριση του γάμου μεταξύ ομοφύλων ε, και η αναγνώριση της εταιρική ε, σχέσης μεταξύ ομοφύλων. Είναι θέμα πολύ σημαντικό αλλά και πολύ ευαίσθητο. Πιστεύω ότι οι καταστάσεις ε, περιέχουν πολλές αμφισημίες και σίγουρα πολλές διαφορές από χώρα σε χώρα. Όμως, δεν υπάρχει λόγος κατά την άποψή μου να υπάρξει πλήρη συνένεση ας πούμε όσον αφορά τον γάμο μεταξύ ομοφύλων αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής. Να υπάρχουν δηλαδή κάποιες βασικές διασφαλίσεις. Βλέπω με ενδιαφέρον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρότι έχει βικτοριανές ε, ρίζες στην ουσία τώρα τελευταία ε, έχει πολύ προχωρημένη νομοθεσία όσον αφορά τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι είναι απόδειξη του βρετανικού πραγματισμού. Ενώ εμείς στη Γαλλία νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο το ρυθμό μας, έχουμε αργοπορήσει. οι ενώσεις, ε, η συμβίωση μεταξύ ατόμων άλλου φύλου ή ιδίου φύλου που έχουν αναγνωριστεί σε άλλες χώρες αναγνωρίζονται με δυσκολία στην ε, Γαλλία. Και βεβαίως πάντα έχουμε το πρόσκομα του γάμου μεταξύ ομοφύλων. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό δίκαιο. Πραγματικά πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο, όποιο κι αν είναι, ένα λοιπόν ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο θα ενθάρρυνε την αναγνώριση εταιρική σχέση ή σύνδεσης ή γάμου ε, μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ε, που θα αναγνωρίζεται και σε χώρες άλλες από αυτές τις οποίες έχει συναυθεί νομίζω ότι θα είναι ένα ε, καλό πρώτο βήμα και δεν μπορούμε να περάσουμε ένα τέτοιο μήνυμα στις υψηλές αρχές που εσείς αντιπροσωπεύετε εδώ. Και με τον τρόπο αυτό να έχουμε ελπίδα ότι θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Σίγουρα Η Γαλλία βρίσκεται ε, μεταξύ των χωρών που έχουν ήδη ανοίξει την πόρτα. Δεν, λέω, δεν αναφέρομαι σε αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν πλήρη απαγόρευση αυτών των σχέσεων, αλλά η Γαλλία είναι από τις χώρες που έχει ανοίξει την πόρτα και νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να την ανοίξει τελείως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γερουσιαστά. Συγκεκριμένε ερωτήσει τέθηκα προ την κυρία Μπέκερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω. Καταρχήν, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει κυρωθεί ακόμη, δεν ισχύει ακόμη και γι' αυτό είναι πολύ νωρί να κάνουμε έναν απολογισμό επ' αυτού. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επιλεγεί ε, το καθεστώ αυτό για να συλλέξουμε εμπειρίε, αλλά ακόμη υπάρχουν υπάρχουν αμφιβολίες διότι έχει θυγεί ένα ευαίσθητο σημείο. Πρόκειται για ένα θέμα με το οποίο ε, μπορεί κανείς να ελέγξει περισσότερο αυτές τις διασυνοριακές σχέσεις και υπάρχουν και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν στη συμφωνία αυτή ε, και ε, από ό,τι ξέρω η ε, Γερμανίδα και η Γαλλίδα η υπουργό δικαιοσύνη έχουν ε, αποστείλει επιστολή προς τους ομολόγους τους των άλλων κρατών για να προσχωρήσουν δηλαδή να μην είναι μία ταχύτητα των δύο κρατών αλλά των 6, 8, 10 ίσως και περισσότερων που θα προσχωρήσουν στη συνθήκη αυτή. Έχω και εγώ την ίδια αίσθηση με εσάς κυρία Μπέκερ ότι βρισκόμαστε σε μία φάση που πρέπει να την περάσουμε μέχρι να φτάσουμε σε συμφωνία σε επίπεδο 27 ή ακόμη περισσότερο χώρο μετά τη διεύρυνση. Μιλάμε για δύσκολα και πολύ λεπτά ζητήματα οικογενειακού δικαίου που τελικά επαφίονται στη διακριτική ευχέρεια και στις χειρονομίες των κρατών μελών. Από ευρωπαϊκή άποψη, εμείς μπορούμε να επικεντρωθούμε στις, στους τομείς όπου έχουμε εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η απόπειρα επίλυσης πολύ ευαίσθητων ζητημάτων για ορισμένες χώρες όπως είναι η σχέση μεταξύ, ε, η γάμη μεταξύ ομοφιλοφίλων, το θέμα υιοθεσίας κτλ. Είναι θέματα όλα αυτά που μπορούμε πρώτα απ' όλα να το λύσουμε με διμερείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες πολύ πιο σύντομα από ό,τι αν περιμέναμε να καταλήξουμε σε πανευρωπαϊκή συμφωνία. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εμπειρία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση για καλές συμφωνίες και λύσεις. Μια και δεν έχω άλλους ε, επίδοξους ομιλητές, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον γερουσιαστή, στον κύριο Αρκάντιο Δία για να μας κάνει μια ανακεφαλαίωση του, των θεμάτων αυτού του πάνελ. Έχετε το λόγο κύριε Γερουσιαστά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για ένα θέμα πολύ απτό και ουσιαστικό για την ε, ευρωπαϊκή καθημερινότητα. Έχουμε δύο ανθρώπους, διαθρώπινα όντα, ενήλικα, όρημα, που καταλήγουν σε συμφωνία για το πώς θα ρυθμίσουν τη συμβίωσή τους. Υπάρχει ένα θέμα επί της ουσίας, αν θα πρέπει το κράτος ε, να κυδεμονεύσει, να αναγνωρίσει, να δώσει νομική υπόσταση ή ένομες συνέπειες σε μια προσωπική απόφαση που αφορά την ιδιωτική ζωή δύο ανθρώπων. Αυτό συζητούμε χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά εργαλεία που δεν είναι εμπειρικά, αλλά είναι αξιολογικά. Γι' αυτό το λόγο τόσοι πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη ζούμε από το δίκαιο, γιατί είναι μια αξιολογική επιστήμη το δίκαιο, δεν είναι μια εμπειρική επιστήμη. Και αν προσθέσουμε και το γεγονό ότι έχουμε την ιδιωτική σφαίρα, έχουμε την ε, ατομική ελευθερία, και το γεγονός ότι οι κοινωνιολόγοι λένε ότι έχουμε τουλάχιστον 17 οικογενειακά πρότυπα ή μοντέλα, με όλο αυτό το συνδυασμό βλέπουμε ότι πραγματικά είναι τεράστια η περιπλοκότητα του σημερινού ζητήματος. Και από ακαδημαϊκή άποψη και από πανεπιστημιακή άποψη το θέμα είναι δύσκολο. Έχουμε μία φοβερή περιπλοκότητα. Είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε με απλό τρόπο κάτι περίπλοκο. Και α μην περιμένουμε απλέ απαντήσει για κάτι που είναι εκφίσω περίπλοκο. Δεν υπάρχουν απλέ απαντήσει για τα περίπλοκα θέματα. Και οι πανεπιστημιακοί πολύ σωστά μα έδειξαν όλο αυτό το φάσμα τη περιπλοκότητα που αντιμετωπίζουμε. Στι πρώτε παρεμβάσει ακούσαμε πολιτικού ηθήνοντε. Εκεί είχαμε πιο γενικέ παρατηρήσει. Οι πανεπιστημιακοί επέμειναν στην περιπλοκότητα της σημερινής κατάστασης και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο ε, μας παρουσίασαν και ένα διμερή τρόπο προσέγγιση αυτού του θέματος, όπως συνέβη στην Γαλλογερμανική Συμφωνία. Νομίζω ότι η εμπειρία αυτή είναι σημαντική και θα πρέπει να μείνουμε στα θετικά της στοιχεία. Για την κατάσταση των πραγμάτων γνωρίζαμε από πριν την περιπλοκότητα. Αλλά ακούγοντα όλε αυτέ τι παρατηρήσει, συνειδητοποιούμε περισσότερο και το βάθο και την πυκνότητα και την περιπλοκότητα και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν διμερεί πρότυπα και υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι νομικής αναγνώρισης ε, με βάση το χαρακτηρισμό της προέλευσης μιας ένωσης. Επίσης μας προτείνεται αναγνώριση και σεβασμός της νομοθεσίας άλλων χωρών γιατί αυτό είναι ένα πολιτιστικό βήμα, ένα πολιτιστικό άρμα, μια πρόοδος και μια πολιτιστική κατάκτηση. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε αυτή την αναγνώριση. Βρισκόμαστε στα τέλη του 2010. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ξεκινώντας από αυτή την πολυμορφία, από αυτή την περιπλοκότητα, αυτή την ανάγκη αναγνώρισης των εθνικών νομοθεσιών, γιατί και το δίκαιο είναι ένα πολιτιστικό επίτευγμα, μια πολιτιστική κατάκτηση που την υλοποιήσαμε μέσα σε 21 αιώνε, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την ανελικτική πορεία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την πρόοδο. Όσοι προτιμούν τη διμερή λύση, καλώς να το πράξουν. Όσοι προτιμούν την λύση μεταξύ 14 χωρών, μπράβο τους. Το ιδεώδες, και εδώ ε, θα μείνω σε μια χειρονομία που έκανε, σε μια χειρονομία που έκανε ο πρόεδρος, γιατί ε, όταν είπε κάποιο ότι καλό θα ήταν να συνεργαστούν 27 χώρε, ο πρόεδρο κουνούσε το κεφάλι του συγκαταβατικά. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτή τη γλώσσα του σώματο του πρόεδρου, που είναι ένα έξω, ένας εξολεκτικό τρόπο επικοινωνία, να πω ότι μπορούμε και 27 να κατευθυνθούμε προ ένα κοινό στόχο. Να δικαιώσουμε του μισθού μα. Γιατί ο μόνο ε, λόγο που δικαιώ, μα δικαιώνει, που δικαιολογεί του μισθού που λαμβάνουμε, είναι να είμαστε χρήσιμοι προς τους συμπολίτες μας. Εγώ ως δικαστής πάντρεψα και χώρισα πολλά διαφορετικά ζευγάρια. Ο πόνος όμως, η οδύνη είναι ίδια στο διαζύγιο. Αλλά και η χαρά των γονιών είναι ίδια. αν, άσχετα με το, τη σύνθεση του ζευγαριού. Αν λοιπόν ε, γίνουμε πιο χρήσιμοι σήμερα, επειδή θα διδαχθούμε ένα από τον άλλον, αν καταφέρουμε να συνεχίσουμε την πρόοδο, ποια και είναι η μορφή, τότε δεν θα έχουμε χάσει το χρόνο μα, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμη και υποφελή αυτή η παρουσία μα εδώ στι Βρυξέλλε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά. Είναι περιττό να προσθέσω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις και την ανακεφαλαίωση που είχατε την ευγενική είναι να κάνατε. Να προχωρήσουμε λοιπόν με έξυπνο τρόπο αντικειμενικό και πρακτικό. Γιατί μερικέ φορέ χρησιμοποιούμε αρχικά Ρώμη 3, Βρυξέλλε 1, βρυξελλε 2 2α. Όλα αυτά είναι ακατανόητα για του ευρωπαίου πολίτε. Ο πολίτη ενδιαφέρεται για την ουσία, για το περιεχόμενο, γιατί προβλέπουν οι νομοθετικέ διατάξει και πώς τον εξυπηρετούν. Συμφωνώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε σαφείς και ξεκάθαρου ορισμού και για το οικογενειακό δίκαιο. Για να μιλούμε με το ίδιο επίπεδο κατανόησης και έτσι πραγματικά να οικοδομήσουμε το κοινοτικό μας δίκαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους πανελίστες γιατί πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, εμπεριστατωμένες, μεστές και πανέξυπνες ε, οι παρεμβάσεις και νομίζω θα αποτελέσουν ε, σημαντικό βοήθημα και στις ε, βουλευτικές και στις δικές μας εργασίες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Ντιές Τεχέρα, την Γραμματεία και μια και έφτασε η 12η μεσημβρινή, θα σας πρότεινα να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της Συνόδου που αφορά τις διασυνοριακές ε, κληρονομιές και διαθήκες. Θα ήθελα να καλέσω εδώ τον Κουρτ Λέχνερ, τον μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για να προεδρεύσει και τον Λόρδο ε, Μπράουνες της Βουλής των Λόρδων. Να σας προσκαλέσω στο Προεδρείο και να σας ευχαριστήσω θερμά.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 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως σας είπα, μόλις είπα ότι θα μπορούσα να έχω κάνει την εισαγωγή και από τη θέση μου και να παραμείνει ο κύριος Τσβίφκα εδώ. Αλλά εάν έτσι συνηθίζετε, τι να κάνω, υποκλίνομαι. Ε, θέλω να χαιρετήσω αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να είναι αποδοτική η συζήτηση, διότι εν αντιθέσει με την Βρυξέλλες 1, Βρυξέλλες 2, Ρώμη 1, Ρώμη 2, τις, ε, ε, τα νομοθετήματα στο στο ιδιωτικό δίκαιο. Πρόκειται για ένα νέο κανονισμό ο οποίος μας δημιουργεί κάτι τελείως καινούριο. Επιπλέον και αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα και ενδιαφέρει και τη συζήτηση γι' αυτό έχουμε εδώ τους εθνικούς βουλευτές πρέπει να μην, να μην θίξει ε, τα άλλα δίκαια. Υπάρχουν όμως επικαλύψεις και είναι αναπόφευκτο να θυγούν και τα δίκαια άλλων θεμάτων. Οπότε, ήθελα να σας πω ότι έχουμε 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν σε μία χώρα άλλη από την πατρίδα τους και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό θανάτων με διασυνοριακές επιπτώσεις και θα αναφέρω εδώ μόνο ένα παράδειγμα. Εάν ένας Πολωνός και Γερμανός, και, και ε, ένας Γερμανός υπήκος ζουν στη Γαλλία ή στο Βέλγιο και έχει περιουσιακά στοιχεία ε, στη Γαλλία ή στο Βέλγιο και στην Πολωνία ή στη Γερμανία τότε από πολωνικής και γερμανικής απόψεως θεωρείται ότι η κληρονομία πρέπει και για τη Γαλλία και για το Βέλγιο να γίνει αναλόγως στην Πολωνία σαν πολωνική κληρονομιά και στην Γερμανία σαν γερμανική και πρέπει εδώ να σας πω ότι έκανε ένα λάθος για το Βέλγιο δεν ισχύει αυτό μόνο από, γερμανι από γαλλικής πλευράς μάλλον αντίστροφα ένας Γάλλος και ένας Βέλγος υπήκος έχουν τελειώσει τελευταία διαμονή στη Γερμανία ή στην Πολωνία. Οπότε στην Γαλλία η κληρονομιά ρυθμίζεται σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο ενώ εις το Βέλγιο σύμφωνα με την τελευταία, τον τελευταίο τόπο του διαμονής διότι το θέμα αυτό ρυθμίζεται διαφορετικά και δεν υπάρχει δυνατότητα να συγκλίνουν οι αποφάσεις και θα πρέπει ε, το θέμα να ρυθμιστεί ε, δικαστικά διότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διαφοροποιούνται. Ορισμένοι βασίζονται στην υπηκότητα, άλλοι στον τελευταίο τόπο διαμονής με πολλές ε, διαφορές και πολλές αποκλήσεις. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και ε, αν χρησιμοποιήσουν το ίδιο δίκαιο και οι δύο διάδικοι θα μπορεί εις ε, το ένα κράτος να αναγνωριστεί η απόφαση αυτή και στο άλλο όχι. Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα εναρμόνισης όπως επρόκειτο για τα προηγούμενα θέματα τα οποία επεξεργαστήκαμε ούτε για μία εφαρμογή όσο προς τα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας όπου υπάρχει μία σύγκληση μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού δικαίου χωρίς να χρειαστεί να ισχύσει για όλους. Θα ήθελα να σας πω ότι επίσης είναι πολύ ε, πρέπει να αποδοθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα των μεταφράσεων διότι αν το κείμενο γαλλικό μπορεί στις μεταφράσεις να προκύψουν φοβε... Ε, σημαντικά προβλήματα. Ως προς την ουσία της προτάσεως πρέπει να σας πω ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι το εφαρμοστέο δίκαιο και το αρμόδιο δικαστήριο στο μέλλον ε, θα πρέπει να ε, βασιστεί είτε στο, στη συνήθη ε, διαμονή του αποθανόντος ή να ε, δέχεται να παραβλέψει αυτό το, ε, ε, αυτό το στοιχείο. Οπότε το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να είναι ο τελευταίος τόπος διαμονής αλλά πρέπει να επιλέξει ο, ο, αποθανόν κατά την διαθήκη του αυτό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει ένα δίκαιο υπό αυτά σας προϋποθέσεις. Πρέπει ε, να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και των διαφόρων εγγράφων. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα πιστοποιητικό θα τα, αυτά μια συμβολιογραφική πράξη, πράγματα τα οποία θα θίξει ο κύριος Δεπασκάλης. Υπάρχει το θέμα του εφαρμοστεί δικαίου που θα θίξει ο κύριος Ζέγκ και ε, το πιστοποιητικό διαδοχής που θα θίξει ε, η κυρία Λέγκα Λεσέη. Πρέπει να σας πω ότι από αυτή τη βάση μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε ή στη συζήτηση για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χρόνο μας ε, διότι υπάρχουν πολλά λεπτομερή θέματα που θα φυγούν και εγώ θα αναφερθώ μόνο επιγραμματικά στα πιο βασικά. Καταρχήν πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο αλλά το ουσιαστικό δίκαιο ενδέχεται να παρουσιάσει ε, ε, επικαλύψεις ε, όσον αφορά το κληρονομικό καθεστών και την κατανομή της ε, ε, ε, των κληρονομουμένων. Υπάρχουν πολλές φορές πολλά προβλήματα τα οποία δεν είναι θέμα των συμβολογραφικών πράξεων αλλά θέμα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου δικαίου και πολλές φορές λέμε αν θα πρέπει να, να καθορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε συνήθις τόπος ε, διαμονής αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να περιληφθεί ένας τέτοιος ορισμός στα κείμενα ε, διότι σε περισσότερα νομοθετήματα τα οποία έχουμε σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει μία τέτοια μνήα. Επειδή είναι πολύ σημαντικό θα ήθελα να αναφερθώ στο, άρθρο 27 του Order Public που αναφέρεται εις ε, τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στα εθνικά κοινοβούλια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και ε, εδώ ε, βλέπουμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ συγκινησιακό και εγώ το ίδιο είχα το πρόβλημα και όταν το εξέτασα λεπτομερώς είδα ότι έχουμε υπερτιμήσει το θέμα αυτό διότι σε όλα τα κράτη-μέρη υπάρχει δυνατότητα ε, και σε αυτό θα μας τα πει και ο συνάδελφος από την το Ενωμένο Βασίλειο όπου δεν υπάρχει ε, δίκαιο καταγεγραμμένο αλλά αποφασίζει ο δικαστής. Πρέπει να σας πω ότι τα προβλήματα τα οποία θα θυγούν ε, ισχύουν ήδη. Ε, έχουμε μία απόφαση του, της Βελγικής Γερουσίας η οποία κατακρίνει μία απόφαση δικαστική και υπάρχει και το θέμα της ε, μετάφρασης. Δηλαδή, οι Βέλγοι ε, εάν, εάν έχουν μετικήσει δεν υπόκεινται πλέον ε, το βέλγικο κληρονομικό δίκαιο και πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ε, αν ε, με τικήσει ε, κάποιος σε ένα άλλο κράτος δεν επαρκεί να επιλέξει αυτό το κράτος σαν ρύθμιση της κληρονομιάς σου πρέπει να πεθάνει εκεί. Οπότε και αυτό είναι κάπως πιο περίπλοκο αλλά δεν θα αποτελέσει το ουσιαστικό αντικείμενο αντικείμενο της συνεδριάσεώς μας όπου θέλουμε να αναφερθούμε περισσότερο στις κοινωνικές πτυχές του θέματος. Όσον αφορά τα έγγραφα, όπως σας είπα, ε, ο κύριος Πασκάλης θα τα σχολιάσει ε, και στη συνέχεια ο Μέτρ Σασά ε, το θέμα του εφαρμοστέου δικαίου και της προστασίας των μελών της οικογένειας. Πρέπει να σας πω όμως ότι ορισμένες διατυπώσεις είναι λανθασμένες και θα έπρεπε να προσαρμοστούν. Ε, ίσως με μια ε, αιτιολογική ε, παραγραφό διότι ε, ήδη στο αρχικό κείμενο δεν ε, είναι σωστή η διατύπωση και χειροτερεύει στις μεταφράσεις. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό διαδοχής θα το αναφέρει κύριος Λεζέ και θα ήθελα να σας πω τι είναι αυτό το πιστοποιητικό το οποίο δεν υπάρχει παντού ε, σε όλα τα κράτη. Είναι η τελεσίδικη απόφαση του, του δικαστηρίου, δηλαδή μια δικαστική πράξη ε, και πρέπει να ε, διαφοροποιήσει κανείς την εφαρμογή στην ουσία με την εφαρμογή της δικαστικής ε, αποφάσεως. Διότι δηλαδή, τουλάχιστον στη Γερμανία ε, η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπάρχει ε, μία απόδειξη διαδοχής και γενικώ η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στη Γερμανία χωρίς να αποτελεί το ουσιαστικό αποδεικτικό στοιχείο εάν, εάν όμως κάποιος διασυνοριακά θέλει να κληρονομήσει κάτι μπορεί να χρησιμοποιήσει το ε, πιστοποιητικό το οποίο μόλις ανέφερα ε, και ε, πιστεύω ότι γι' αυτό αυτό το πιστοποιητικό περί της Διαθήκης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε διασυνοριακές ε, περιπτώσεις διότι ε, το, το θέμα δεν μπορεί να ρυθμιστεί παντού ικανοποιητικά διότι ο καθένας ξεκινά από, τη δικιά του, από τις δικές του προϋποθέσεις υπάρχουν διαφορές υπάρχουν προβλήματα τα οποία ισχύουν ακόμη και αν μειώνονται σιγά σιγά διότι με τον κανονισμό αυτό περί των κληρομη, νομιτηρίων ε, έχουμε μία καλύτερη απεικόνηση της θέλησης του αποβιώνοντος και της αποδείξης ε, όπου ισχύει αυτό το θέμα. Οπότε ε, δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα διότι ε, όσοι ζουν, συνεχίζουν να ζουν ή στην ε, χώρα, ε, στη χώρα τους δεν, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και η περιουσία τους στο εξωτερικό βελτιώνεται διότι έχουν περισσότερα δικαιώματα σύμφωνα με το νέο αυτό κανονισμό. Βέβαια και στο Συμβούλιο είναι ακόμη δύσκολη κατάσταση διότι ε, το θέμα είναι περίπλοκο και ελπίζω ότι θα είναι αίσια η έκβαση του διότι πέρυσι είχα υποβάλει ένα έγγραφο είναι όμως και θέμα γοήτρου για τα κράτη-μέλη υπάρχουν νέα στοιχεία και γι' αυτό ελπίζω ότι στην αρχή του επομένου έτους Bildung, Entschuldigung, einen Berichtsvorschlag vorlegen werde, äh, damit dann im και θα υποβάλω ένα έγγραφο το οποίο μπορεί να βοηθήσει ίσως στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και σας δίνω τον λόγο. Äh, Bitte um Entschuldigung, Herr Pascalis. Ja, darf ich Sie bitten? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι με το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, για το δίκαιο διαδοχής ο κοινοτικός νομοθέτης έχει πλέον μια μεγάλη ευκαιρία να παρέμβει σε ένα τομέα ενδεχομένως περιορισμένο που όμως αφορά ε, εκ του συνεγγύς και πολύ συχνά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ε, ε, αναφέρομαι στην χρήση δημοσίων εγγράφων στις διαδικασίες διαδοχής. Κυρίως πρόκειται βεβαίως για συμβολεογραφικές πράξεις αλλά και έγγραφα άλλου είδους από άλλες δημόσιες αρχές. Είναι προφανές ε, σε περιπτώσεις διαδοχής λόγω θανάτου ε, χρειάζονται οπωσδήποτε τέτοια δημόσια έγγραφα. Επί παραδείγματι μπορούμε να δώσουμε το αντίγραφο της Διαθήκης, ε, την κοινοποίηση, δημοσιοποίηση, την αποδοχή ή αποποίηση της Διαθήκης, ε, την καταγραφή των αγαθών, την ρευστοποίηση ή παραχώρηση, καθώς επίσης και την διανομή ε, της ε, ε, διαδοχής. Αυτό που θέλουμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε με το σχέδιο κανονισμού το οποίο συζητάτε είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να ε, χρησιμοποιεί ή να προσφεύγει σε ε, κάποιο δημόσιο έγγραφο συχνά ε, πρόκειται επαναλαμβάνω για συμβολιογραφική πράξη ενώπιον του συμβολιογράφου της δικής του χώρας που θα μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία θέλουμε να επιτρέψουμε να δώσουμε την δυνατότητα δυνατότητα στις αρχές μιας χώρας ε, να χρησιμοποιήσουν ένα ε, δημόσιο έγγραφο το οποίο προέρχεται από άλλη χώρα σαν ε, απολύτως αποδεκτό υποκατάστατο αντιστοίχου εθνικού εγγράφου. Γιατί λοιπόν αυτή η δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης τέτοιων εγγράφων θεωρείται σημαντική και χρήσιμη και για τον πολίτη και για, τον, για τις αρχές, μα για λόγο, για τον απλό λόγο ότι το δημόσιο αυτό έγγραφο χρησιμοποιείται ε, για λόγους ε, σαν ασφαλής ε, τεκμηρίωση έτσι ώστε να αποτελέσει πιστοποιημένο έγγραφο και να, να δίνει την κατεξοχή τη δυνατότητα χρήσης σαν αποδεκτικού στοιχείου και λόγω του περιεχομένου και λόγω των δηλώσεων που σε αυτό περιέχονται. Θα ήταν κρίμα λοιπόν αυτού του είδους ε, η ε, νομική βεβαιότητα που δίνεται μέσα από αυτού του είδους τα έγγραφα ε, να χάνεται όταν το έγγραφο χρησιμοποιείται σε χώρα άλλη από αυτήν στην οποία έχει εκδοθεί. Απέναντι στην ε, ανάγκη ε, ελεύθερης χρήσης ε, και αναγνώρισης αυτών των εγγράφων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε αυτή την περίπτωση οι ισχύουσες σε κάθε χώρα διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Βεβαίως μπορεί να διαφέρουν ε, οι διατάξει ή μπορεί να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται διαφορετικά από τις διοικητικέ ή ε, δικαστικές αρχές της εν λόγω χώρας που είναι διαφορετικές από αυτές που καλούνται ε, να εκτελέσουν τη διαδοχή. στο προσχέδιο το, το, η Παύλα 26 και τα άρθρα 34 και 35 προβλέπουν σαφώς ε, σημαντικούς κανόνες για τη διαστηριακή χρήση των πιστοποιημένων δημοσίων εγγράφων. Η παρουσία αυτών των ε, κανόνων έχει ήδη δώσει λαβή για επικρίσεις και συζητήσεις ε, μέχρι και έτοιμα πλήρους κατάργησής τους. Αλλά κατά την άποψή μου αυτό απορρέει από ενδεχόμενη ελλειπή κατανόηση των ε, ε, άρθρων αυτών οι επικρίσεις ε, λένε ας πούμε ότι δεν κατανοούμε καλά για ποιες πράξεις ε, ε, πρόκειται αλλά σας έδωσα προηγουμένως κάποια παραδείγματα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές για ποιου είδους έγγραφα μιλάμε και ο καθένας από τους παριστάμενους λόγω της προσωπικής του εμπειρίας γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα έγγραφα τα οποία συνήθως εμπλέκονται σε διαδικασίες διαδοχής. Οι επικρίσεις επίσης αναφέρουν ότι δεν γίνεται κατανοητή η αξία που μπορεί να έχουν αυτού του είδους τα έγγραφα ε, στην, ε, ε, στις πρακτικές διαδοχής. Υπογραμμίζουν δε κυρίως ότι δεν θα μπορεί η χρήση τους να εξομοιωθεί με δικαστικές αποφάσεις γιατί φυσικά αυτού του είδους τα δημόσια έγγραφα μπορούν να αμφισβητηθούν ενώπιον δικαστορίων. Αυτό, αυτό είναι προφανές και φυσιολογικό και τέτοιου είδους επικρίσεις ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτοί που τις διατυπώνουν δεν γνωρίζουν καν το περιεχόμενο και την δυνατότητα χρήσης αυτών των ε, εγγράφων που βεβαίως μπορεί να αμφισβητηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ε, αλλά που η ίδια η ύπαρξή τους μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική, πραγματική ε, στην χώρα στην οποία έχει εκδοθεί αλλά το ζητούμενο είναι να μπορεί να αναγνωριστεί η αυθεντικότητά τους ε, ε, και σε άλλες χώρες να αναγνωριστεί δηλαδή ότι πρόκειται για επίσημο δημόσιο έγγραφο και στη χώρα έκδοσης αλλά και στην χώρα χρήσης. και βεβαίως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμφισβήτησης ε, αυτού του εγγράφου. Αλλά ε, η δυνατότητα αμφισβήτησης με κανένα τρόπο ε, δεν ακυρώνει το βάρος αυτού του εγγράφου. Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ακόμα κανόνες ε, οι οποίοι ε, να ε, διασφαλίζουν την χρήση, την δυνατότητα χρήση των εγγράφων αυτών και σε άλλες χώρες από τις χώρες έκδοσής τους. Ή μάλλον θα διορθώσω αμέσως λέγοντας ότι δεν είναι αρκετές έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρους χρήσης αυτών των εγγράφων. Πρέπει να δημιουργηθούν λοιπόν αυτοί οι κανόνες που θα διευκολύνουν την χρήση και την ελεύθερη διακίνηση αυτών των ε, πιστοποιημένων δημοσίων εγγράφων. Ήδη το πρώτο στοιχείο που ε, υπάρχει στο κοινοτικό κεκτημένο ε, είναι η αναγνώριση της εκτελεστικής ισχύω που έχουν ε, τα δημόσια έγγραφα και που ήδη περιέχονται στο άρθρο 50 της Συνθήκης των Βρυξελών της 27 Σεπτεμβρίου 1968 όσον αφορά την δικαιοδοσία, την νομική δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση των νομικών αποφάσεων όσον αφορά το εμπορικό και το αστικό δίκαιο. Ε, πράγμα που επιβεβαιώνεται και στον κανονισμό 44 2001 που είναι γνωστό ως Βρυξέλλες 1 που αντικατέστησε την ε, ε, προαναφερθήσα συνθήκη καθώς επίσης επιβεβαιώνεται και από τους άλλους κανονισμούς 2201 κάθετος 2003 και 805 2004 και ακόμα καλύτερα στον, τελευταίο κανονισμό 805 κάθετος 2004 και τον κανονισμό 4 του 2009 όσον αφορά τις υποχρεώσεις διατροφής όσον αφορά ε, τις ε, χώρες civil law που είναι δηλαδή η συμβολιογραφική πράξη εγγράφεται ήδη ε, στο κοινοτικό δικαϊκό σύστημα και έχει και εκτελεστική ισχύ. Επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο υφίσταται στο κοινοτικό δίκαιο είναι η αναγνώριση του δημοσίου εγγράφου ε, έτσι όπως καθορίζεται στην ουσιαστική απόφαση Unibank της 17ης Ιουνίου 1999 ε, ε, πινάκιο 260 97 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η αυθεντικότητα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από δημόσια αρχή θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στο σύνολο του περιεχομένου και όχι μονάχα σε στοιχεία όπω η υπογραφή και επίση ότι το έγγραφο θα πρέπει να είναι εκτελεστέο στο κράτο το οποίο έχει συνταχθεί ε, και ε, στι ε, υπόλοιπε χώρε. Επομένως, Επομένως ε, ε, η αρχή επιβεβαιώνεται ε, και όσον αφορά τον κανονισμό 805 του 2004 και στον κανονισμό 4 του 2009. Και επομένως είναι ένα δίκαιο το οποίο υπάρχει ήδη, αν αναφερθούμε ήδη στις Βρυξέλλες 1 εδώ και 40 χρόνια. Αυτό που λείπει όμως είναι ένας σαφής κοινοτικός κανόνας ο οποίος θα αναφέρεται στην αποδεικτική αποτελεσματικότητα. Ε, και κυρίως όταν αναφερόμαστε στο δίκαιο διαδοχής. Επί παραδείγματι, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, έναν κατάλογο κληρονομητηρίου που θα πρέπει να υπάρχει σαν έγγραφο, ε, σαν ένα πιστοποιημένο δημόσιο έγγραφο και το οποίο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε όλον τον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο έτσι ώστε να αποδειχθεί το δικαίωμα ε, διαδοχής δεν πρέπει να ξεχνάμε επίση ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί ε, με το θέμα αυτό των πιστοποιημένων δημοσίων εγγράφων ε, κάνοντας ε, μία μελέτη των υφισταμένων κανόνων στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να αναφερθώ ας πούμε πρώτα απ' όλα στη μελέτη για την νομιμοποίηση και την δυνατότητα αποστήλε ε, που ε, διενεργήθηκε το 2007 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου Study on the Use of Public Documents in the EU ε, έτσι, όπου αναφέρεται ότι χρειάζεται επιπλέον πιστοποίηση προέλευσης για την αυθεντικότητα του εγγράφου που θα πρέπει να δοθεί από τον συγγραφέα του εγγράφου μια άλλη μελέτη, η οποία κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι η μελέτη την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβολιογράφων σε συνεργασία με την Deutsche Notar Institut ε, και που πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη των δημοσίων εγγράφων σε έξι χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Πολωνία, την Ρουμανία και την Ελβετία ε, από όπου απορρέουν σημαντικά ε, στοιχεία, κυρίως όσον αφορά την διαφορετικότητα ε, των υποεξέταση νομικών συστημάτων. Το Κοινοβούλιο επίσης εκπώνησε και ψήφισε ψήφισμα που ενεκρίθη στο Στρασβούργο την 18η Δεκεμβρίου του 2008 ε, με τίτλο «Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, το, ε, για, την πιστοποιημένη, για το πιστοποιημένο ευρωπαϊκό έγγραφο» με εισηγητή τον κύριο Μανουέλ Μεδίνα Ορτέγα. Νομίζω ότι με όλα αυτά ε, αποδεικνύεται ότι το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία ε, των ε, δημοσίων εγγράφων μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός και μπορεί να κωδικοποιήσει στο κοινοτικό δίκαιο τους ε, κανόνες που θέλουν να διευκολύνουν ε, τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Στη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του κανονισμού δόθηκαν κάποιες βασικές αρχές τις οποίες μπορώ να συνοψίσω ως εξής το ε, αυθεντικό δημόσιο έγγραφο το οποίο ε, ε, γίνεται αποδεκτό σε μια χώρα μέλος μπορεί να έχει αποτελέσματα και σε άλλες χώρες μέλη όσον αφορά την αυθεντικότητά του και την αποδεικτική του ισχύ. Το αυθεντικό δημόσιο έγγραφο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλήρες υποκατάστατο αντιστοίχου εγγράφου στην χώρα που δεν είναι η χώρα προέλευσης. Επίσης και η άλλη πλευρά του, του νομίσματος ε, το δημόσιο έγγραφο ε, δεν μπορεί ε, συγγνώμη, το δημόσιο έγγραφο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης και ελέγχου από ε, οποιαδήποτε εθνική δημόσια ε, αρχή, νομική αρχή στην χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω ότι αυτό το ε, σημείο θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Δηλαδή ότι μπορεί να αμφισβητηθεί και στην χώρα στην οποία έχει εκδοθεί και στην χώρα στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει περαιτέρω να συζητηθούν και να αποσαφινιστούν συνεχιστούν. Επίσης είναι ε, σαφές ότι αυτή η πράξη δεν μπορεί να έχει στην χώρα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί ε, ε, ισχύ μεγαλύτερη από το αντίστοιχο έγγραφο το οποίο ισχύει στην χώρα χρήσης. Πιστεύω ότι με βάση αυτά που μόλις είπαμε μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σύνολο απλών και σαφών κανόνων που τελικά θα διευκολύνουν την διασυνοριακή χρήση τέτοιων εγγράφων και θα διευρύνουν αποτελεσματικότερα τον δικαστικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ντεπασκάλης για αυτή την λεπτομερή παρουσίαση των ε, συμβολογραφικών εγγράφων στην Ευρώπη ασχέτως από αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σασά από τη Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση του κανονισμού του 2009 προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία νομοθεσία που θα εφαρμόζεται για τις κληρονομιές και ε, να υπάρχει ε, ε, ένα στοιχείο με το οποίο να συνδυάζει κανείς την κατάσταση του αποθανόντος με το χρησιμοποιούμενο δίκαιο. Σύμφωνα λοιπόν με της ε, διατάξεις του ε, Ευρωπαϊκής Συμβολιογραφικής Νομοθεσίας ε, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο γερουσιαστής Ιούγκ ότι το δικαίωμα της οικογενείας βασίζεται σε τον πολιτισμό κάθε κράτους. Θέλω εδώ να αναφερθώ στην ρήξη και εις ε, τα προβλήματα της, ε, του ενίου εφαρμοστέου δικαίου και τι περιμένουμε από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Σε ορισμένες χώρες χώρες. Ε, υπάρχει ένα σύστημα όπου διαχωρίζεται η κατάσταση μεταξύ των κινητών και των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και θα πρέπει αυτός ο διαχωρισμός να εγκαταλειφθεί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την κληρονομία των ατόμων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς, πράγμα που έχει τονιστεί και να μην υπάρχουν ε, ρυθμίσεις βάσει διαφορετικών νομοθεσιών, να μην υπάρχει ρευστοποίηση και θα επανέλθω στα, ε, ε, διάφορα χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά επηρεάζεται το οικογενειακό δίκαιο της οικογενείας και αποδυναμώνεται η κληρονομική διαδοχή διότι πολλές πολλές φορές αν υπάρχει επιφύλαξη χρησιμοποιείται ο χώρος όπου βρίσκεται το, το, κληρονομούμενο αντικείμενο ενώ αυτό το στοιχείο δεν ισχύει πάντοτε. Θέλαμε λοιπόν στο άρθρο 27 ε, ο νομοθέτης ε, να ε, διευκρινίσει το θέμα αυτό που ήταν ασαφές για τους χειριστές του και αυτό ίσχυε και για το γαλλικό κοινοβούλιο. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρχει ένα εξαιρετικός χαρακτήρας σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ορισμό της δημοσίας τάξεως και της αρχής της επικουρικότητος. Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε το αποτέλεσμα της ρήξεως αυτής στα πλαίσια του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και της μελλοντικής ασφαλή ασφαλείας των ε, ε, οικογενειακών αλλαγών και ε, των ρυθμίσεων των των κληρονομικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν διαφορετικές λοιπόν απόψεις στα διάφορα θέματα. Καταρχήν όσον αφορά την προστασία της οικογένειας, μία βασική ε, κριτική όσον αφορά ε, το κληρονομικό δίκαιο αναφέρεται στη δυσκολία κάποιος να οργανώσει την διαδοχή του διότι εάν υπάρχουν ακίνητα σε μία χώρα ε, υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση και δεν μπορεί κανείς να ρυθμίσει στους δικαιούχους κληρονόμους την εφαρμογή αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσει κανείς ε, να, ε, ε, να εφαρμόσει ένα σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλους τους ενδιαφερόμενους και θα καλύπτει συγχρόνως και τις διατάξεις δημοσίας τάξεως κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον. Παραδείγματος χάρη, για τη Γαλλία υπάρχει η ε, ε, ε, πρόορη αποποίηση κληρονομίας η οποία εφαρμόζεται τελευταίο στη Γαλλία. Αλλά για να είμαστε ικανοποιημένοι με τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι στα πλαίσια της οργανώσεως της κληρονομίας ότι θα ισχύσει μία μόνο, ένα μόνο δίκαιο και Πρόκειται για διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου που δεν διατηρείται σε όλα τα εθνικά δίκαια σύμφωνα με την πρόταση του 2009 στο άρθρο 17 στη Γαλλία όπου ε, ισχύει το ενιαίο δίκαιο για να προστατευτεί η οικογένεια και το άτομα στο κληρονομικό δίκαιο. Για να εφαρμοστεί λοιπόν αυτή η διάταξη θα μπορεί ο καθένας να ε, αποφασίσει το δίκαιο το οποίο θα ρυθμίσει την κληρονομιά του αλλά λαμβάνοντας υπόψη διατάξεις που δεν θα μπορούσαν να κυρώσουν αυτές ε, τις προθέσεις και να προστατεύσουν την οικογένεια χάρη στον προγραμματισμό της ε, ρυθμίσεως για το μέλλον. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ε, το περιβάλλον και η εγγύτης προς ε, τον αποθανόντα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην τελευταία του, στον τελευταίο τόπο διανομής του θα υπάρχουν ε, και τα, και τα προσωπικά του αντικείμενα και ο τραπεζικός του λογαριασμός, η σύνταξή του και ε, τα περισσότερα ακίνητα εφόσον αυτά θα περιλαμβάνουν και την ε, κυρία ε, διαμονή που αποτελούν τα στοιχεία της κληρονομιάς και μόνο βάσει αυτών μπορεί κανείς να πει ίσως ενδιαφερομένους ότι μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αποθανόντος. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η εγγύτης προς την, ε, τον τελευταίο τόπο διανομής για να εντομίζονται τα ε, πιο άμεσα στοιχεία του ενεργητικού και της περιουσίας τους κατά τρόπον ώστε ε, να εφαρμοστεί ο νόμος ή το κράτος στο οποίο βρίσκονται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Οπότε είτε η διαδοχή θα γίνει προς τους άμεσους κληρονόμους είτε θα ρυθμιστεί ε, δια του κληρονομικού δικαίου. Υπάρχει η ενιαία ε, ρύθμιση η οποία προβλέπει μία πιο εύκολη ε, ρύθμιση διότι θα μπορέσει καλύτερα έτσι να προστατευτεί η οικογένεια και να υπάρξει σωστή εκτέλεση που θα βασίζεται και στους έμπειρους συμβολιογράφους. Κατά αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν οι ασάφειες και οι οικογένειες θα μπορέσουν να έχουν ένα επιπλέον προσόν από την ε, εναρμόνιση της ε, κληρονομιάς και θα πρέπει το συγκεκριμένο δίκαιο να ε, ε, ρυθμίσει ε, τα διάφορα επιμέρους θέματα όπως παραδείγματος χάρη το δίκαιο της χώρας όπου εφαρμόζεται η ε, κληρονομιά ε, και ε, να διευκρινιστούν διάφορα θέματα που στο παρελθόν δεν υπήρχε εναρμόνιση και για να καταλήξω αν θέλουμε να κοιτάξουμε τις προκλήσεις του κληρονομικού δικαίου για τα μέλη της οικογενείας του απαθανόντος ε, κρυβόμαστε κάπως πίσω από την νομοθεσία και δεν πρέπει να αφήσουμε ε, τις ε, καταστάσεις να ξεφύγουν και να αποφύγουμε να ισχύσει ένα σωστό δίκαιο και θεωρούμε ότι ο τελευταίος τρόπος διαμονής του αποθανόντος είναι ένα στοιχείο άμεσο και ασφαλές για την οικογένεια κατά τρόπον ώστε και οι διάφοροι εμπλεκόμενοι να μπορέσουν να καλυφθούν μέσω των συνήθων αρμοδίων όπως οι συμβολεογράφοι και ε, τέλος τονίζω το, ε, ε, τον λόγο υπάρξεως μιας τυπικής διαδικασίας αναφερόμενο στα σχόλια του καθηγητού Γκριμάλτη του Πανεπιστημίου του Παρισιού όπου ελέγχθη ότι πρέπει να υπάρχει μια τυπική διαδικασία για να αποφύγουμε τις συγκινησιακές καταστάσεις που ξεπερνούν πολλές φορές τη λογική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σασάν για αυτή την εκτενή παρουσίαση του πρόγραμμα της οικογενείας των συγγενών και του τελευταίου τόπου διαμονής και την θετική αξιολόγησή σας και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Λέγκα Λεσάη με συγχωρείτε την κυρία ναι, ε, Λένκα από την Τσεχία να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Λένκα Λεσάη. Όχι Λεσάη, Λεσάη. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, μια μικρή διόρθωση. Θέμα της εισήγησής μου είναι το περιεχόμενο και οι συνέπειες του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα θέμα που θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ολόκληρες, αλλά δυστυχώς έχω μόνο ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή μου και θα προσπαθήσω μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο να αναφερθώ στα ουσιώδη σημεία αυτής της πρότασης. Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο ή Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διαδοχής είναι ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έχετε ακούσει ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουμε πολύ διαφορετικό τρόπο τα θέματα κληρονομικής διαδοχής και αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα δικαιώματα και των εμπλεκομένων μερών. Γι' αυτό και είναι σχεδόν αδύνατον να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για διασυνοριακά ζητήματα. Με το Ευρωπαϊκό Αυτοκληρονομητήριο, με το Ευρωπαϊκό Αυτοπιστοποιητικό Κληρονομικής Διαδοχής θα έχουμε ένα εργαλείο που θα επιτρέπει το ίδιο περιεχόμενο και τις ίδιες συνέπειες και αποτελέσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, άσχετα με το κράτος μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα, τα πιστοποιητικά θάνατος, διαδοχή κτλ. Αυτό προβλέπει το άρθρο 37 της πρώτης κανονισμού ότι στόχος του κληρονομητηρίου, του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου είναι να, χορηγήσει μία απόδειξη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην πράξη της διαδοχής και να διευκρινίσει, να διαλευκάνει την κατάσταση. Λαμβάνεται υπόψη και το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα και οι συνέπειες και γι' αυτό ακριβώς η Ισπανική Προεδρία συνέταξε έναν ορισμό στον οποίο επεσήμανε ότι αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο κρατός μέλος και το άρθρο 36.1 προβλέπει στο κείμενο την πρόταση της ε, Ισπανικής που αισθανίστηκε και η Βελική Προεδρία ώστε να τεθεί σε ισχύ από το 2010 αυτό το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο. Τι περιλαμβάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό. Προβλέπει ότι το περιεχόμενό του θα σταθμίζει τα δικαιώματα των δικαιούχων, των, κληρονο, των κληρονόμων και να λαμβάνει υπόψη και το εύρος των κληρονομούμενων αγαθών θα πρέπει να είναι σαφές το περιεχόμενο αυτού του πιστοποιητικού. Επίσης αυτό το επιστοποιητικό θα πρέπει να είναι απλό και διαφανές και να περιλαμβάνει στοιχεία που με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2. Είναι αναμφίβολο ότι αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία των ε, αρμόδιων αρχών, των αρχών έκδοσης, στοιχεία για τους κληρονόμους, για το εφαρμοστέο δίκαιο στη συγκεκριμένη κληρονομική διαδοχή, πληροφορίες για τα νομικά πρόσωπα και ούτω καθεξής. Μερικά από τα στοιχεία αυτά που προτείνονται χρήζουν ε, ιδιαίτερης προσοχής. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, για παράδειγμα, που αναφέρονται στα σημεία A, G και K. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Αυτοπιστοποιητικό δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες αυτές του H, ε και ι. Υπάρχουν ε, ορισμένες διατάξεις που προβλέπουν ε, διανομή της κληρονομίας μεταξύ των κληρονόμων. Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν στο στόχο του πιστοποιητικού. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τον κατάλογο, την απογραφή των κληρονομούμενων αγαθών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εδώ διαφορές. Το πιστοποιητικό αυτό δεν πρέπει να προβαίνει σε ένα κατάλογο των δικαιωμάτων των κληρονόμων, ούτε να περιορίζει αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπουν τα σημεία ΙΤΑ και Ε. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού. Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό επίσης δεν αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία δικαιωμάτων κληρονομίας. Το πιστοποιητικό αυτό αναφέρεται μόνο στην, εθνική, στην εφαρμοστή εθνική νομοθεσία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και για την πληροφορία αυτή θα πρέπει να ανατρέξουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο. Αυτό θα βοηθήσει για την άντληση συγκεκριμένων πληροφοριών. Ούτε θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό να είναι ένας κατάλογος δράσεων που θα πρέπει να γίνουν από τον εκτελεστή της Διαθήκης στο διαχειριστή τον κληρονόμο. Ποια λοιπόν θα πρέπει να είναι τα αποτελέσματα, οι ένομε συνέπειε αυτού του Ευρωπαϊκού Κληρονομιδίου. Με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται ταυτόχρονα αυτόματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί γίνεται λόγος για δικαστικές αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα αναφέρεται και σε ποιες περιπτώσεις δεν λαμβάνεται υπόψη η δικαστική απόφαση. Η ορολογία που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό προβλέπει εξασφάλιση των δικαιωμάτων και των συνεπειών της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων όπως ε, πρότεινε και η Ισπανική Προεδρία, αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα πρέπει να προκαλεί ένα με σε όλα τα κρατημέλη χωρίς ε, περαιτέρω διαδικασία. Θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξει του εδαφείου 2 της παραγράφου 32 και γι' αυτό να θεσπίζονται και διάφορα εχέγγυα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 34 38 και 43. Οι δικονομικές αυτές εγγυήσει μας δίνουν μια πολύ καλή βάση και δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για αυτές τις ε, δικονομικές εγγύσεις. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι για να έχει ένομε συνέπειε αυτό το πιστοποιητικό, αυτό το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πάσει στιγμή διακρύβωση του κύρου του, τη εγκυρότητά του. Ή να διαπιστωθεί αν έγιναν κάποιε αλλαγέ σε ό,τι αφορά το βασικό περιεχόμενο του κληρονομητήριου. Από αυτή την άποψη ήταν χρήσιμο και ένα ηλεκτρονικό μητρό, όπω προβλέπει και η έκθεση του Ινστιτούτου Max Planck είναι να ότι ένα τέτοιο ηλεκτρονικό μητρό θα ήταν πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε περίπτωση τεκμηρίου κληρονομικών δικαιωμάτων για συγκεκριμένα είδη κληρονομικής διαδοχής. Είναι κάπως προβληματικό το θέμα της προστασίας της α, καλής πίστης, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4. Αυτή η προστασία της καλής πίστης είναι κάτι που επαφίεται στις αρμόδιες αρχές. Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε και τις διατάξεις ε, του, της παραγράφου 5 της, Ευρω... της του παραρτήματος 5 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει ότι το πιστοποιητικό αυτό θα ισχύσει και για τα εθνικά μετρό. Βέβαια, δεν μπορεί να αποτελεί αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό από μόνο του νομική πράξη δεσμευτική θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που εμπίπτουν στο κοινό δίκαιο, για παρά, όπως αναγνώρισε και το Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό κληρονομίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο κράτος για λόγους κληρονομικής διαδοχής και θα πρέπει να συνδυάζεται, παραλαμβάνω, και με άλλα έγγραφα. Γιατί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκυρο έγγραφο μόνο εφόσον το απαιτήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ευχαριστώ κυρία Λεσάη για αυτή την παρουσίαση του περίπλου ο, θέματος που δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη και τώρα έχω διάφορους που ζητούν το λόγο. Έχουμε 10 λεπτά χρόνο. Ο κύριος Τομέη έχει ζητήσει το λόγο από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση ε, ότι εφόσον εγώ βρίσκομαι εδώ πρέπει να σας πω ότι είμαι κάπως επιφυλακτικός για ορισμένα θέματα. Δηλαδή αν θέλει κάποιος ένα τέτοιο πιστοποιητικό το οποίο ελπίζουμε ότι θα ισχύσει και θα εφαρμοστεί πρέπει να ισχύσει και το νομοθέτημα οπότε πρέπει να σας πω ότι ε, προς το παρόν είμαι επιφυλεκτικός κατά δεύτερον λόγο θα ήθελα να σας πω ότι έχω ορισμένε επιφυλάξεις σχετικά με ε, ε, την, το, έγγραφο δημοσιοποίησης αλλά βεβαίως ε, πρέπει να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε σαν ε, στοιχείο εάν θα είναι ο τόπος τελευταίας διαμονής ή την υπηκότητα και ε, εξαρτάται από το δίκαιο διαδοχής το οποίο διαφέρει αναλόγως των χωρών από τις παρατηρήσεις όμως της κυρίας Λεσάη διαπίστωσα ότι το θέμα του καταλόγου θα, αύριο θα συζητήσουμε το θέμα του καταστατικού όπου εγγράφονται ε, όλα αυτά τα έγγραφα και ίσως το βιβλίο το όπου αναφέρονται ε, οι άδειε διαμονής είναι το κατάλληλο έγγραφο. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο αυτά θέματα. Ευχαριστώ Κύριο Γιόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια παρατήρηση στο θέμα του κληρονομητηρίου. Πριν από μερικούς μήνες ε, στη Γαλλική Γερουσία συζητήσαμε το θέμα αυτό και βεβαίως ε, μετά από ε, την κοινοτική πρωτοβουλία εμείς αντιδράσαμε θετικά. Όμως επιστήσαμε την προσοχή και της γαλλικής κυβέρνησης και των διαφόρων ευρωπαϊκών αρχών επί του γεγονότος ότι στη Γαλλία και ίσως και σε άλλες χώρες, δεν το γνωρίζω, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος ονομάζεται ε, κληρονομική, ε, κληρονομικό αποθεματικό ή ε, κληρονομικό αποθεματικό, βάσει του οποίου 2 τρίτα, 1 τέταρτο, 1 πέμπτο, ανάλογα με τα παιδιά, ανάλογα με τους κληρονόμους, έχουν τη δυνατότητα να βάλουν σε αποθεματικό ένα τμήμα της κληρονομιάς για να το χρησιμοποιήσουν αργότερα. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή των νομοθετών το γεγονός της ύπαρξης αυτού του μηχανισμού ε, γιατί στη Γαλλία είναι ιδιαίτερος προσφυλής ε, αυτή η διαδικασία και ε, είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα πρέπει λοιπόν να αντικατοπτρίζεται και αυτή η πραγματικότητα στον νέο κανονισμό. Κάποιος ίσως θα μπορούσε να μας ενημερώσει για το πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίες για το θέμα αυτό. Äh, Τότε και εγώ θα ήθελα σύντομα να σχολιάσω. Δεν θέλω να κατακρίνω το Γερμανικό Κοινοβούλιο, αλλά αναφέρθηκα και στη γερουσία του Βελγίου. Είναι καλό να, ε, να εξετάζει κανείς ε, ε, τους νομοθέτες ε, που ασχολούνται με αυτό το θέμα και πολιτικά θα πω ότι τους λυπάμαι που το αναλαμβάνουν και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι πριν 5-6 χρονών όταν συζητούσαμε την πράσινη βίβλο τα συναισθήματά μου ήταν σαν τα δικά σας και αφού ασχολήθηκα με το θέμα ενδελεχώς διαπίστωσα ότι αν έχουμε δικαίωμα επιλογή είναι ε, σωστό και μόνο έτσι μπορεί να ρυθμίσει. Δηλαδή το θέμα της υπηκότητος, ε, εάν το επιβάλλουμε ε, δεν έχετε δικαίωμα επιλογής και ξέρετε ότι πρέπει να έχετε επιλογή, δηλαδή για να μείνετε κάπου πρέπει να έχετε ήδη διαμείνει εκεί επί τρία χρόνια ή κάτι άλλο. Μόνο με τέτοιους συνδυασμούς ο συνήθους χώρου διαμονής με δικαίωμα επιλογής μπορώ να δεχθώ και να ερμηνεύσω αυτή τη ρύθμιση. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητάμε διεξοδικά είναι ότι στην προηγούμενη ε, τελευταία κοινή συνέλευση οι συγητές είχαν συζητήσει με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Υπουργών και ε, ένα Γάλλο καθηγητή από το Παρίσι, τον καθηγητή Μπερτό, ο οποίος είχε κάνει μία μελέτη επί του θέματος και πρέπει να το θυμόμαστε. Πρέπει επίσης να σας πω ότι αν ε, ε, κοιτάξτε ε, την ρύθμιση και τους συνδυασμούς δεν αλλάζουν τόσα πολλά στοιχεία. Πολλά στοιχεία παραμένουν κοινά διότι ένας Γερμανός υπήκος ο οποίος ζει στη Γαλλία, έχει παντρευτεί μια Γαλλία και έχει, Γαλλίδα και έχει μείνει εκεί πολύ καιρό εάν ε, ε, ε, τα μετακινηθεί και ε, καταθέσει τα χρήματά του στη Γερμανία και μεταφέρει και την έδρα του στην Γερμανία τότε δεν, δεν μπορεί η Γαλλία να κάνει τίποτα διότι η διαδοχή θα ρυθμιστεί σύμφωνα με την ε, γερμανική νομοθεσία αλλά όχι ακριβώς διότι εντωμεταξύ έχει αλλάξει και η γαλλική νομοθεσία οπότε εάν κοιτάξουμε συλλογικά τις εξελίξεις θα δούμε ότι δεν υπάρχει μια ουσιαστική επιδείνωση και ε, δεν φύγονται τα τα δικαιώματα όσων δεν ε, διακινούνται διασυνοριακά. Απλώς θελήσαμε να υπάρξει μία ρύθμιση το οποίο να καταλήξει στην έκβαση την οποία επιθυμούσαμε. Και τώρα δίνω το λόγο ε, τον Ρόδο για ε, τα τελικά σχόλιά του. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Επιτροπή σας για τη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης. Βέβαια και εμένα με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και όπως και εσείς γνωρίζω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ασθενίζεται αυτή τη στιγμή ούτε συνυπέγραψε αυτές τις προτάσεις. Και μάλιστα σε αυτό επιδοκιμάστηκε και από την Επιτροπή στην οποία προεδρεύω στη Βουλή των Λόρδων. Εξετάσαμε την πρόταση της Επιτροπής με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια και επισημάναμε πολλές περιπλοκότητες, πολλές δυσκολίες που τις ακούσαμε και σήμερα το πρωί. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ο ίδιος ο πρόεδρος, αλλά και ο συνάδελφός σας από την Bundestag ε, επισήμαναν αυτές τις δυσκολίες θέλω κι εγώ να γίνω ένα παράδειγμα του χαρακτηριστικού εγγλέζου που μας περιέγραψε ο κύριος Χάιντελ το πρωί. Διαπιστώνουμε την ανάγκη αλλαγή, διαπιστώνουμε και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες όταν υπάρχουν διασυνοριακά θέματα κληρονομικής διαδοχής, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι στην προσπάθεια να υιοθετήσουμε μια γενική λύση που θα τα καλύπτει όλα, ελοχεύει ο κίνδυνος ε, ανεπιθύμητων συνεπειών και περαιτέρω περιπλοκή σε ορισμένους ε, άρα επιδείνωση τη κατάστασης. Και μάλιστα η δράση στα θέματα αυτά έχει τόσο άμεση σχέση με τα εθνικά δίκαια και τις εθνικές διατάξεις για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν νομίζω ότι έχει νόημα μια πανευρωπαϊκή λύση. Το ίδιο συνέβη και για τα ποινικά θέματα. Εκεί είχαμε σημαντική επιτυχία και πολύ σταδιακά με συγκεκριμένα βήματα και όχι από μια γενική πρόταση που θα τα καλύπτει όλα. Βέβαια, όντως παραδέχομαι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ίσως έχει άλλα προβλήματα περισσότερα, περισσότερα νομικά προβλήματα από άλλε χώρες εξαιτία της νομικής τους παράδοσης με τα θέματα κληρονομιάς και περιουσιακών στοιχείων, αλλά πιστεύουμε ότι ο διαθέτης ε, είναι ε, ελεύθερος να διαθέσει την περιουσία του όπως θέλει. Ούτε υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα σε μας. Και θα ήθελα να σας ζητήσω λίγη κατανόηση ο ρόλος των συμβολογράφων είναι ιδιαίτερος στο Ηνωμένο Βασίλειο και σας μιλάω γιατί έχω πείρα από το επάγγελμα αυτό. Είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά των συμβολογράφων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαφορετικά σε άλλες χώρες. Δεν είναι η ε, ίδια η αξία που έχει η συμβολογραφική πράξη σε όλες τις χώρες και σίγουρα δεν είναι ισοδύναμη με μια δικαστική πράξη, μια δικαστική απόφαση. Και έτσι έρχομαι στο πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου, Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Κληρονομικής Διαδοχής. Ήταν τόσο γενική η πρόταση όταν την εξετάσαμε, ώστε περιλάμβανε όχι μόνο δικαστικές αποφάσεις, αλλά και συμβολογραφικά πιστοποιητικά, συμβολογραφικέ πράξεις. Αρκεί κάτι τέτοιο για να δικαιολογηθεί η μετάθεση, μεταφορά μιας ε, περιουσιακών στοιχείων από ένα κράτος σε άλλο, χωρίς τα δέοντα εχέγγυα που περιμένουμε. Επίσης, το πρόβλημα έχουμε με τα, έγγραφα, τα δημόσια έγγραφα ή τα έγγραφα δημοσιοποίησης. Βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο συγγνώμη, παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη, εξέλιξη αυτής της πρότασης. Αυτό είναι βέβαιο. Και δεν θα ήθελα να καταλήξω σε συμπέρασμα για το αν είναι δόκιμο να εμείνουμε στην ε, αποχή μας ή να το προσυπογράψουμε. Πάντως το θέμα της συνήθως κατοικίας ως ε, συνδετικός κρίκος για το καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου χρήζει περαιτέρω λεπτομεριών και τελειοποίησης. Θέλουμε να διευρυνθεί η δυνατότητα και να καλύπτεται περισσότερο η ελεύθερη επιλογή του διαθέτη. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε και το δικαίωμα φόρου κληρονομιά και τη ε, ίσπραξης του φόρου κληρονομιά από το αρμόδιο κράτος. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Η απολούσευση της διαδικασίας και η διατήρηση των ειδικών κληρονομικών καθεστώτων είναι αντίφαση από μόνη της. Ανησυχητικές και οι δυνατότητες ανάκλησης το θέμα της εφαρμογής των δημοσίων εγγράφων επίσης είναι επίμαχο. Δυστυχώς δεν μπορώ να συμπαραταχθώ με τους συναδέλφους από άλλες χώρες. Αν ήμουν πιο νέος και μόλις ε, ε, άρχισε την άσκηση του συμβολογραφικού επαγγέλματο, θα ήμουν πολύ πιο ενθουσιώδης με τις προτάσεις σας, γιατί είναι πολύ πιο επικερδές να μπορεί κανείς να είναι ε, συμβολογράφος σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είχαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για προβληματισμό και νομίζω ότι όλοι οι εθνικοί βουλευτέ θα ήθελαν να εντρυφήσουν σε αυτό το θέμα πολύ πιο λεπτομεριακά πριν καταλήξουμε σε ένα οριστικό συμπέρασμα. Πάντως, ε, εγώ και λόγω τη Νομική παράδοσης θα προτιμούσα η χώρα μου να ενταχθεί σε αυτή την πρόταση παρά να κρατήσει αυτοεξαίρεση. Πάντως είναι τόσο περίπλοκο το θέμα που θα προτιμούσα μια πιο σταδιακή ε, λύση βήμα προς βήμα από ότι μια γενική λύση που θα καλύπτει τα πάντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λόρντ Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι σύμφωνα με τους Βρετανούς συναδέλφους ε, το θέμα αυτό συζητείται και στο Ενωμένο Βασίλειο και θα δούμε στο τέλος εάν θα ε, ε, συμπορευτεί και το, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήξερα ότι εις, ε, το, ε, την Αγγλία δεν υπάρχει γραπτό δίκαιο αλλά εφόσον είμαι πολιτικός διαπίστωσα ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και ήδη ε, έχουμε κοινά στοιχεία σε κάτι που είπε στην πρώτη του φράση Λόρδος για τη φορολογία διότι ουσιαστικά αυτό που εννοούσε δεν ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό που καταλαβαίναμε εμείς γι' αυτό σας το επισημαίνω διότι πολύ εύκολο είναι να, να υπάρξουν παρανοήσεις αλλά βάσει της πρωτοβουλίας μας η Επιτροπή ε, ξεκίνησε ε, ε, μία συζήτηση επί επί της φορολογίας όχι για να υπάρχει ε, ενιαία ε, φορολογική αντιμετώπιση αλλά ε, για να υπάρχει κάποια σύγκληση διότι δεν υπάρχουν σε πολλές χώρες συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας και πολλές φορές υπάρχει φορολογικό θέμα και για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες σε πολλές χώρες. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το θέμα δεν είναι κάτι που θα επιλύσουν ούτε οι νομικοί ούτε οι πολιτικοί αλλά το λέγω εις της ε, τις ε, εκπροσώπους των χωρών όπου ισχύει ε, το καθεστώς της ε, ε, εγκαταστάσεων και σε ορισμένες χώρες ε, υποχρεούνται τα δικαστήρια να χρησιμοποιήσουν τον νόμο της Σαρία. Τώρα τουλάχιστον αυτό θα καταργηθεί με την πρόοδο αυτή η οποία θα επιτευχθεί και όπου επί δεκαετίες ή και εκατονταετίες ίσχυε το θέμα της υπηκότητος. Γι' αυτό και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ε, υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία και ιδίως η ελευθερία επιλογής του χώρου διαμονής, ε, της χώρας διαμονής. Ε, ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν, όσους παρενέβησαν, όσους άκουσαν προσεκτικά. Ολοκληρώνουμε την πρώτη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα.